Ας αρχίσουμε την απογευματινή συνεδρίασή μας, αγαπητοί συνάδελφοι. Να καλωσορίσω θερμά εκ μέρου σας την Εσθονική Προεδρία και τον Υπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα της Προεδρίας, ο οποίος και θα είναι και ο πιο προβεβλημένος ε, άνθρωπος. Έχουμε τον κύριο Μάσικας, που είναι επιφορτισμένος και με διαπραγματεύσεις στον τομέα αρμοδιότητάς μας. Γι' αυτό είναι μαζί μας. Σας συγχαίρω. Να σας πω ότι εδώ στο Κοινοβούλιο πολύ συχνά βλέπουμε ότι οι προεδρίες που ασκούνται από μικρές χώρες πολύ συχνά είναι πολύ αποτελεσματικές και δεν φίδονται προσπαθειών για την προώθηση του προγράμματός τους. Ε, ελπίζω ότι σαν Εστονική Προεδρία θα είσαστε φημισμένοι για την ψηφιακή διάσταση της ζωής μας και θα προωθήσετε το όλο θέμα. Ο κ. Χαουρέγκη ε, είχε επεξεργαστεί την ψηφιακή δημοκρατία και συζητήσαμε το θέμα και ήρθαν εμπειρογνώμονε εδώ και στον εμπειρογνώμονε ήρθαν εδώ και συζητήσαμε τον εκλογικό νόμο, εκλογές μέσω διαδικτύου, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρα ξέρουμε τις πρακτικές που ακολουθείτε όσον αφορά τα ψηφιακά. Θέλουμε να ακούσουμε τις προτεραιότητές σας και κυρίως εκείνες που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας. Λοιπόν, χωρίς να χρονοτριβήσουμε, να σας δώσουμε το λόγο, κύριε Υπουργέ, για να μοιραστείτε μαζί μας τα θέματα που αφορούσαν την Προεδρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει ο κύριος Υπουργός, κυρία Πρόεδρε, μεγάλη τιμή για μένα να παρίσταμε εδώ η Ιστονική Προεδρία εκτιμά πολύ την συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα πρέπει να πω προσωπικά εκτιμά την καλή συνεργασία με την Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων συνεργασία που ήδη ξεκίνησε εδώ και ένα δίμηνο και ήδη διεξήχθησαν καρποφόρες ανταλλαγές απόψεων επί αρκετών ζητημάτων κοινού μας ενδιαφέροντος. Η Προεδρία μας, όπως σωστά αναφέρατε, κυρία Πρόεδρε, είχε, ήρθε έξι μήνες νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί, λόγω του Brexit και αυτό τονίζει ε, την ε, κατάσταση που επικρατεί γεμάτη ε, αναταράξει το ΣΥΠΗΝ, το κλίμα όταν ξεκινήσαμε το σχεδιασμό της Προεδρίας μας το 2012, εκεί είχαμε την κρίση ε, της Ευρωζώνης που συγκλώνησε το κοινό νόμισμα της Ένωσης μετά από δύο χρόνια περίπου είχαμε τη μεταναστευτική κρίση που πόρα απέχει από το να περάσει και εκτίθεται η Ένωση σε αυτό το πρόβλημα στηρίχθηκε η νομοθετική διαδικασία που έπρεπε να αντιμετωπίσει μια πάρα πολύ δύσκολη κρίση από πλευρά επιχειρησιακή και οι συνέπειε αυτή τη κρίση είναι ακόμα αισθητέ σήμερα. Σήμερα πιστεύω ότι η κατάσταση στην Ένωση είναι κάπως διαφορετική και το κλίμα στην Ένωση είναι κάπως διαφορετικό από ό,τι πριν από ένα χρόνο μετά από το δημοψήφισμα για το Brexit. Έχουμε ξανά ανάπτυξη οικονομίας. Η υποστήριξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Τα 27 κράτη-μέλη μπόρεσαν να συμφωνήσουν στην Βρατισλάβα, στις διακηρύξεις στην Πρατισλάβα και της Ρώμης επί της μελλοντικής κατευθύνσεως της ε, Ενώσης αλλά το βασικό μάθημα που αποκομίσαμε και ακόμα μαθαίνουμε από αυτές τις κρίσεις είναι η προηγηθήσα και συνεχιζόμενη κρίση. Ότι πρέπει να ξαναποκτηθεί η νομιμότητα της Ένωσης στα μάτια των πολιτών. Εκείνα που θεωρούσαμε σαν δεδομένα, τα στοιχεία αυτά, δεν είναι πλέον κάτι δεδομένο. Η νομιμότητα της Ένωσης πρέπει να κατακτηθεί εκ νέου και καθημερινά να καταβληθεί αυτή η προσπάθεια. Πρέπει να συνεχίσουμε την δουλειά μας αναπτύσσοντας περαιτέρω το όλο θεσμικό σύστημα της Ενώσεως. Ταυτοχρόνως πιστεύουμε ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για ανάκτηση της νομιμότητας είναι να πετύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και να δώσουμε συγκεκριμένα ωφέλη στους πολίτες μας. Για εκείνους οικοδομούμε και συντηρούμε την Ένωση. Αυτός λοιπόν είναι ο ακρογωνίος λήθος. Αυτή είναι η βασική αρχή της Εστονικής Προεδρίας. Να πετύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα για τους πολίτες μας. καθορίζοντας τις προτεραιότητες της ε, Προεδρίας μας, και επεξεργαζόμενοι τις συμφωνίες που θα οδηγήσουν στα ωφέλη για τους πολίτες, εμείς έχουμε εστιαστεί επί τεσσάρων βασικών τομέων προτεραιοτήτων. Καταρχάς, ανοιχτή και καινοτόμα ευρωπαϊκή οικονομία. Δεύτερον, ασφαλή Ευρώπη. Τρίτον, ψηφιακή Ευρώπη, ελεύθερη διακίνηση δεδομένων. Τέταρτον, μία βιώσιμη Ευρώπη για όλους. Αυτές οι προτεραιότητες λαμβάνουν υπόψη τα βασικά στοιχεία όπως το στατηγικό θεματολόγιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η διοργανική συμφωνία, οι νομοθετικές ε, προτεραιότητες. Βέβαια, οι αποφάσεις της Μπρατισλάβα και της Ρώμης, των συνόδων κορυφής σε αυτές τις δύο πόλεις, αναφέρονται σε αυτά. Να αναφέρω ακροθυγώς τους βασικούς στόχους στους τέσσερις τομείς προτεραιοτήτων και μετά θα αναφερθώ στα ζητήματα και τα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν ε, αυτή την επιτροπή. Ανοιχτή και καινοτόμω ευρωπαϊκή οικονομία. Τι σημαίνει, Να δημιουργήσουμε καλύτερε ευκαιρίε για τι επιχειρήσει και του πολίτε, να προωθήσουμε τι θέσει εργασία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να απελευθερώσουμε γι' αυτό το πλήρε δυναμικό τη ενιαία αγορά. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει όλο το δυναμικό τη ενιαία αγορά. Το μεγαλύτερο μέρο τη δυναμικότητα δεν, δεν το έχουμε αντιλήσει πρέπει να δημιουργήσουμε ένα προβλέψιμο επιχειρησιακό περιβάλλον, τραπεζικό τομέα και να, έχουμε, να αυξήσουμε επίσης τις διαπραγματεύσεις για, με εμπορικό περιεχόμενο και να κάνουμε βήματα προς καθαρότερη ενέργεια. Για την ασφαλή ε, Ευρώπη, η ασφάλεια είναι κάτι που περιμένουν περισσότερο από όλα οι Ευρωπαίοι πολίτες από την Ευρώπη, η τρομοκρατία, την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο, η προστασία εξωτερικών συνόρων, τα σημαντικά θέματα. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα γεγονότα εκτό των συνόρων. Οι συνεχιζόμενε συζητήσει για αυτά τα θέματα καταδεικνύουν ότι χωρί μια κοινή αντίληψη είναι δυσχερέστατο να έχουμε αποτελεσματικέ λύσει. Η Εστονική Προεδρία βασίζεται κατά πολύ στο καλό έργο της Μαλτέζικης Προεδρίας επί πολλών θεμάτων. Αντιμετωπίζουμε την αστευτική κρίση και αντιμετωπίζουμε και το δυσχερέστατο πρόβλημα της αλληλεγγύης στα πλαίσια της αναθερήσεως του κοινού συστήματος ασύλου και του κανονισμού του Δουβλίνου. Η τρίτη προτεραιότητά μας είναι η ψηφιακή Ευρώπη και η ελεύθερη ε, διακίνηση στοιχείων, δεδομένων. Η προετοιμασία του εδάφους για πραγματική ψηφιακή ε, Ευρώπη είναι διτή διαδικασία. Επεξεργαζόμεθα καταρχάς τα χαρτοφυλάκια τη ενιαία ψυχική αγοράς μέσω νομοθετικών προτάσεων, να σταματήσει ο γεωγραφικό αποκλεισμό καλύτερες ε, υπηρεσίε, καλύτερο κανονισμό όσον αφορά τι ηλεκτρονικέ επικοινωνίε κλπ. Και απελευθέρωση των μέσων επικοινωνία Ταυτόχρονα έχουμε σαν στόχο να δρομολογήσουμε συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί των βαθιών αλλαγών που δημιουργούνται από, το ψηφιακή, από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και αλλαγές που θα γίνουν σε όλους του τομεί τη ζωής λόγω αυτής της μεταμορφώσεως. Συνεχίζεται αυτή η ψηφιακή αλλαγή, επηρεάζονται όλες οι οικονομίες και όλες οι κοινωνίες. Αυτή η συζήτηση είναι κάτι καινούριο για όλους μας. Και πρέπει να γίνει καλύτερα αντιληπτή η προσέγγιση. Χρειάζεται ενδελεχέστερη ανάλυση για να μπορέσουμε σαν Ευρώπη και σαν Ένωση να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεταμόρφωση. Τώρα, το πιο ορατό γεγονός που διοργανώνει στον Στονική Προεδρία είναι η ψηφιακή σύνοδος κορυφής στο Ταλίν στις 29 Σεπτεμβρίου. Θα συμμετάσχει ο πρόεδρος Ταγιάννη και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. η Σύνοδος Κορυφής θα οδηγήσει σε αυτές τις ζητήσεις που ανέφερα. Θα οδηγήσει σε ευαισθητοποίηση για αυτές τις αλλαγές. Και η συζήτηση θα γίνει στο ύψιστο δυνατό επίπεδο. Η προετοιμασία της Σύνοδο Κορυφής είναι σε πρώιμα στάδια ακόμα, αλλά δεν θα με εξέπλησε αν οι τρεις βασικοί τομείς που θα εστιαστούμε θα ήταν πρώτα απ' όλα η κυβερνοασφάλεια, δεύτερον οι ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της μεταμορφώσεως αυτής και τρίτον, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου είναι σημαντικότατη στις συζητήσεις. Η, η έκθεση για την ηλεκτρονική δημοκρατία θετήθηκε φέτος τον Μάρτιο και είναι πολύτιμο εργαλείο συνεισφορά στα πλαίσια του θεματολογίου για την ηλεκτρονική δημοκρατία. Τέταρτος τομέας βιώσιμη Ευρώπη για όλους, να καλύπτονται, να συμπεριλαμβάνονται όλοι. Πρέπει η ποιότητα ζωής να διατηρηθεί στα σωστά επίπεδα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Βλέπουμε πώς η ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών αλλάζει τη φύση της εργασίας. Αυτό ζητεί να προσέξουμε τις συνθήκες εργασίας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ισορροπία εργασίας ιδιωτικής ζωής και επίσης τη χορήγηση ίσων ευκαιριών στην αγορά εργασίας. Και τώρα κυρίες και κύριοι να αναφερθώ στα θέματα που αφορούν την Επιτροπή σας, την Επιτροπή ΑΦΚΟ. Θέλουμε να συνεχίσουμε το έργο των προηγουμένων Προεδριών της Συμβουλίου σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή σας, με τα μέλη της και θέλουμε να προχωρήσουμε στα σημαντικά ζητήματα που έχουν σημασία για όλους μας. Θα ξεκινήσω με την εφαρμογή της Διοργανικής Συμφωνίας για καλύτερη νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια της Εστονικής Προεδρίας κάνουμε αποτίμηση της εφαρμογής αυτής της ε, συμφωνίας. Θα προωθήσουμε περαιτέρω την όλη διεργασία. Ήδη έχουμε κάνει κάποια βήματα σχετικά με αυτό το θέμα. Την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο συμμετείχα σε συνεδρίαση πολιτικού επίπεδου σχετικά με το άρθρο 40 αυτής της Ιρωνικής Συμφωνίας, δηλαδή ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και ήδη ξεκινήσαμε το έργο καθορισμού ημερομηνίας για την επόμενη συζήτηση που θα γίνει σε πολιτικό επίπεδο. Ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες. Οι πρώτοι εμπειρογνώμονες συναντήθηκαν και συζήτησαν το θέμα των κατεξουσοδότησης πράξεων και των εφαρμοστικών πράξεων, κάτι που θέλουμε να προωθήσουμε ως ζήτημα. Αυτές οι συναντήσεις που διεξήχθησαν την πρώτη εβδομάδα της Προεδρίας μας, προετοίμασαν, προελίαναν το έδαφος καθοδόν προς μια συνεδρίαση ε, σε πολιτικό επίπεδο που θα γίνει και θα κάνει μια αποτίμηση των εξελίξεων στο δεύτερο εξάμεινο. Άλλο σημαντικό θέμα είναι το Brexit. Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση νωρίτερα σήμερα αυτή η Επιτροπή ε, έκανε ανταλλαγή απόψεων με τον συντονιστή του Κοινοβουλίου για τον Brexit, τον κύριο Βερχόφστατ. Είναι ύψη της σημασία να διατηρήσουν την ενότητα οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, την ενότητά μας Πρέπει λοιπόν να διατηρηθεί η ενότητά μας στην διαπραγματευτική διαδικασία. Ε, η συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου είναι κρισίμου σημασίας. Και οι διευθετήσεις για αυτή τη συνεργασία, οι ρυθμίσεις για αυτή τη συνεργασία υφίστανται. Δράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πολύτιμη συνεισφορά του στην όλη διαδικασία μέχρι τώρα, κυρίως με το ψήφισμα που υιοθετήθηκε στην Ολομέλεια αρχές Απριλίου. Αυτό μας βοήθησε το Συμβούλιο να παγιώσουμε τις θέσεις μας, να ενοποιήσουμε τις θέσεις μας. Αυτό ε, βοήθησε. Και προσβλέπω στην συνέχιση αυτής της ε, καλής συνεργασίας. Τώρα, εν των ευρωεκλογών του 2019 παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τις συζητήσεις σχετικά με τις προτάσεις του Κοινοβουλίου για την κατανομή των εδρών. Είναι περιπλοκότατο το ζήτημα. Κατανοούμε πολύ καλά τους λόγους για την καθυστέρηση της ε, αντίστοιχης πρότασης. Βέβαια όλοι πρέπει να έχουμε υπόψη ότι για να διεξαχθούν οι εκλογές Εν ευθέτω χρόνο, το 2019, η τελική απόφαση θα πρέπει να υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έγκαιρα. Και έγκαιρα σημαίνει κατά προτίμηση πριν το επόμενο καλοκαίρι για να προλάβουν τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν όλα τα αναγκαία μέτρα Εκτιμούμε ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο ε, έχετε εμπλέξει τα κράτη-μέλη στην ε, προπαρασκευαστική εργασία τα διάφορα σεμινάρια που διοργανώσατε και είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διαβούλευση. Το Μητρό Διαφάνειας είναι μία από τις προτεραιότητές μας για το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Η Μαλτέζικη Προεδρία σημείωσε σταθερή πρόοδο με βάση την πρόταση που έχει υποβληθεί και εμείς ε, δεσμευόμαστε να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο ούτως ώστε να έχουμε μία σαφή θέση όλων των κρατών μελών. Θέλουμε να συνεργαστούμε και με εσά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαστε ανοιχτοί σε συζητήσεις πολιτικού επίπεδου όσο ταχύτερα γίνεται. Για τον εκλογικό νόμο τώρα. Δεν είναι εύκολο θέμα και το λέω με ήπιο τρόπο. Διότι τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές ε, παραδόσεις και ρυθμίσεις και διαφορετικούς εκλογικούς νόμους εκτιμούμε τις προσπάθειες που ανέλαβαν οι δύο τελευταίες προεδρίες, αλλά τελικά οι συζητήσεις απεδείχθησαν πολύ πιο περίπλοκες, ιδιαίτερα για το δικαίωμα των πολιτών να ψηφίζουν σε τρίτες χώρες και για τα ελάχιστα κατόφλια η Προεδρία μας δεσμεύεται να συνεχίσει τις συζητήσεις στα πλαίσια του Συμβουλίου και με την Επιτροπή σας. Και να συζητήσουμε και πώς θα μπορούσαμε να σημειώσουμε πρόοδο σε αυτό το περίπλοκο θέμα. Το δικαίωμα δημιουργίας εξεταστικών επιτροπών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει μια σειρά από περίπλοκα θέματα. Περιμένουμε την έκβαση της διαβούλευσης που διεξάγεται τώρα από τις τρεις νομικές υπηρεσίες. Υπάρχουν και νομικά και θεσμικά θέματα που πρέπει να διευκρινιστούν και ελπίζω το αποτέλεσμα αυτής της νομικής διαβούλευσης να διευκολύνει την επίτευξη πρόοδου. Δεσμευόμεθα να συνεχίσουμε την προσπάθεια και να διερευνήσουμε περαιτέρω δυνατότητες. Το Συμβούλιο έχει επανειλημμένα δεσμευθεί να προωθήσει τις προσπάθειες ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ξέρουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μέσω της γνώμης του, του Δεκεμβρίου 2014 έθεσε μια σειρά από περίπλοκα νομικά θέματα. Η ανάλυση και αντιμετώπιση των θεμάτων η πρόταση μιας μεθόδου για να επιτευχθεί πρόοδος είναι δύσχερης υπόθεση αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο φορέας που θα πρέπει να διαπραγματευτεί την ένταξή μας άρα περιμένουμε την πρόταση της Κομισιόν για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα αναπομένοντα θέματα που έθεσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα δράσουμε περαιτέρω όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάσει την ανάλυση της. Τώρα για τον κανονισμό για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Το Κοινοβούλιο, ε, το Συμβούλιο διόρισε πρόσφατα δύο ε, από τα μέλη της Επιτροπής Διακεκριμένων Ειδικών. Περιμένουμε την αναθεώρηση του υπάρχοντος κανονισμού για να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα που υπάρχουν. Ο οποίος κανονισμός ε, μόλις τον περασμένο Ιανουάριο τέθηκε ενισχύει. Ξέρω ότι σήμερα η Επιτροπή σας θα κάνει μια ανταλλαγή απόψεων για μια ενδεχόμενη θεώρηση. Ω Συμβούλιο είμαστε διατεθειμένοι να εξετάσουμε το ενδεχόμενο θεώρηση εάν η Επιτροπή υποβάλει πρόταση για το θέμα αυτό. Για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών. Συμφωνούμε απόλυτα με το Κοινοβούλιο. για το σημαντικό ρόλο αυτής της δυνατότητας για να προσεγγίσουν οι πολίτες της Ένωσης, αλλά γνωρίζουμε και τις αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος. Οπότε αναμένουμε την πρόταση της Επιτροπής για να αναθεωρηθεί αυτή η πρωτοβουλία, ο κανονισμός αυτός, και μόλις υποβληθεί αυτή η αναθεωρημένη πρόταση, θα αρχίσουμε να το εξετάζουμε. Πολλά θέματα λοιπόν. Πολύ δουλειά λοιπόν χρειάζεται και πολλή αφοσίωση. Εσείς μπορείτε να θεωρείτε το Συμβούλιο ως έναν έντιμο διαμεσολαβητή και αφοσιωμένο εταίρο στην προσπάθειά σας για τα θέματα αυτά αλλά και για άλλα θέματα που ε, έχουν σημασία για τους πολίτες μας. Ευχαριστώ. Δεν χειροκροτούν συχνά οι συνάδελφοι, οπότε τα πήγατε πολύ καλά. Ε, μόνο τέσσερις συνάδελφοι να πάρουν το λόγο, όχι. Α, ξέρω, ξέρω ποιοι έχω ζητήσει το λόγο. Πέντε, ωραία. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να έχουμε ερωταποκρίσεις ε, αλλά όχι πάνω από 5 λεπτά για τον καθένα. Οπότε, αν μπορείτε να περιορίσετε τι ε, ερωτήσει σα στα 2 λεπτά για να απαντάει 3 λεπτά μετά ο κύριο Υπουργό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει ο κύριο Σέφλιν. Και σα καλωσορίζω από πλευρά του ΕΛ και είναι χαρά μα που σα έχουμε εδώ. Εντυπωσιάστηκα από τον τρόπο με τον οποίο ε, παρουσιάσετε τα θέματα. Τρία θέλω να θέσω. Αρχίσατε πολύ σωστά ξεκινώντας για το ότι πρέπει να κερδίσουμε την νομιμοποίησή μας. Να κερδίσουμε και πάλι δηλαδή την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μετά ε, αναφερθήκατε στα ψηφιακά θέματα. Ξέρω ότι η Εστονία είναι πρωτοπόρα σε σχέση με πολλές άλλες χώρες που θα μπορούσα να αναφέρω Πώς συνδέονται αυτά. Κατά τη γνώμη μου, ένα μεγάλο τμήμα της πολιτικής ε, αντιπαράθεσης λαμβάνει χώρα ψηφιακά και οι ψηφιακές δεξιότητες ε, είναι λοιπόν κάτι το οποίο συμβάλλει ιδιαίτερα. Και ξέρω ότι στην Εστονία ήδη υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου. Το έχω διαπιστώσει, δεν είναι απλώς ε, σχέδιο, είναι πραγματικότητα. Δεύτερον, ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων βεβαίως. Ζωτικό αλλά τίθεται και το θέμα της κυβερνοασφάλειας. Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο. Πήγα στο Τάλιν πολύ πρόσφατα σε μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής Πολιτισμού. Θα θυμάστε ότι έκανε πολύ κρύο και το Σαββατοκυριακό. Ναι, αλλά δεν φταίει η Προεδρία για τον καιρό, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριο Σέπλιν, δεν είμαι και τόσο σίγουρος οι Εστονοί θα μπορούσαν να ψηφιοποιήσουν και το κλίμα. Αλλά εντυπωσιάστηκα από την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Εστονία για τα θέματα κυβερνοασφάλειας. Βέβαια δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρχει απόλυτη κυβερνοασφάλεια ποτέ. Άρα πώς επιλύεται τα θέματα αυτά σε συνδυασμό το ένα με το άλλο. Το δεύτερο θέμα είναι η ανακατανομή εδρών. Πολύ δύσκολο. Ξέρετε ότι η θέση του ΕΛΚ είναι, γιατί είμαστε κάπως συντηρητικοί, είναι να μην γίνει καμία αλλαγή, να παραμείνει το status quo, να μην ανακατανεμηθεί καμία από τις έδρες. Αλλά τότε έχουμε το πρόβλημα ότι η Σουηδία και η Ουγγαρία έχουν τον ίδιο αριθμό βουλευτών αλλά η Σουηδία έχει 130.000 πολίτες παραπάνω. Εντάξει δεν είναι τόσο πολύ αλλά κάτι είναι. Η Ουγγαρία αυτή τη στιγμή αν γίνει ανακατανομή θα πάρει 21 έδρες ενώ η Σουηδία θα έχει μόνο 20. Οπότε η λύση να μην υπάρξει καμία ανακατανομή η Σουηδία θα κάνει προσφυγή. Θα στοιχημάτιζα παρά το ότι δεν μου αρέσει να στοιχηματίζω, θα στοιχημάτιζα ότι θα το κάνει. Τι θα γίνει γι' αυτό. Δεύτερον, εγώ θεωρώ την εξή αντίφαση. Η ανακατανομή γίνεται με βάση τον πληθυσμό. Αλλά λόγω των δημογραφικών αλλαγών των τελευταίων 25 ετών που αφορούν και την Εστονία θα το ξέρετε γύρω στα 20 εκατομμύρια πολίτες έχουν μεταναστεύσει από τα κράτη-μέλη της Ανατολικής Ευρώπης. Η Πολωνία, για παράδειγμα. Πολλοί Πολωνοί έχουν φύγει. Αυτές είναι οι επιπτώσεις της ε, ενιαίας αγοράς. Έτσι πρέπει να λειτουργεί. Όλοι αυτοί οι οποίοι μετακινήθηκαν πώς εκπροσωπούνται δεν είναι κάτι που θα επιληθεί το επόμενο εξάμεινο, αλλά θα πρέπει να το έχετε υπόψη. Και αν έχετε καμία πρόταση για το πώς να λυθεί, ίσως και μέσω της ψηφιοποίησης, δεν ξέρω, θα βρω αρπαστικές τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ, Τζόζο, Θα χρησιμοποιήσεις ε, για... για τις ερωτήσεις σου, ενώ όλο τον χρόνο αφήσαμε μόνο 29 δευτερόλεπτα στον Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ όσο συνοπτικότερα γίνεται. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ κύριε Σέπφλη. Να σας τα πω λοιπόν επιγραμματικά. Νομιμότητα, νομιμοποίηση οποιασδήποτε κυβέρνηση ακόμα και της ευρωπαϊκής κυβέρνησης, Την πρώτη στιγμή που θα κάνεις ε, την δήλωσή στη φορολογική online, όπου και αν κάθεσαι, στα πρώτα δύο λεπτά, δηλαδή όπου έχεις σύνδεση με το ίντερνετ, ε, από τη στιγμή που μπαίνεις και το κάνεις έτσι, λατρεύεις το σύστημα. Γιατί το συγκρίνεις με τις δεκάδες σελίδες, τις οποίες έπρεπε να συμπληρώσει χειρόγραφα. Και κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο είναι ένα από ε, μία από τις πολλές υπηρεσίε που σου προσφέρει η κυβέρνηση είναι ακριβώς αυτή η ευκολία. Και τι κάνει αυτό, νομιμοποιεί την κυβέρνηση στα μάτια του πολίτη που διευκολύνεται. Και ασφάλεια βέβαια, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι δεν αποτελεί μυστικό το ότι σε διάφορα κρατημέλη και σε διάφορα κράτη γενικότερα υπάρχουν κυβερνήσεις που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις απειλές προς την κοινωνική ασφάλεια που ε, προέρχονται από διάφορες πηγές. Ε, για κάποιους η τεχνολογία αποτελεί πρόβλημα και για άλλους λύση. Γιατί κάποιοι ξεκινούν με την προστασία του ιδιωτικού βίου, με την προστασία των δεδομένων. Πάντως, τα βασικά στοιχεία για την ελεύθερη κυκλοφορία και ροή των δεδομένων είναι καταρχήν να δούμε το θέμα της ιδιοκτησίας αυτής της, ε, αυτών των δεδομένων. Ποιος έχει την κατοχή βεβαίω το άτομο το οποίο αφορούν τα στοιχεία αυτά. Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεχνολογίες που επιτρέπουν μία πιο ασφαλή ροή δεδομένων. Έχουμε το blockchain, ας πούμε, στην Εστονία, το οποίο το χρησιμοποιούμε και αν θέλετε αυτή την εμπειρία μπορούμε να τη μοιραστούμε μαζί σας. Αλλά βέβαια έχετε απόλυτο δίκιο, είναι πολύ στενά συνδεδεμένες αυτές οι δύο έννοιες και θα πρέπει να βρούμε εκείνη τη λεπτή ισορροπία που είναι απαραίτητη. Για την τρίτη σας ερώτηση δεν έχω κάτι παραπάνω να προσφέρω. Όλοι γνωρίζουμε τι πρέπει να γίνει ε, μέχρι τις επόμενες εκλογές και μάλλον έχετε δίκιο. Γιατί αντιμετωπίζετε το θέμα με πολύ ρεαλισμό. Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να τα καταφέρουμε και αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή καθήμενος σε τούτη εδώ την καρέκλα. Μπρέσο, παρακαλώ, τρία λεπτά όμως, όχι παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω Ιταλικά. Αν θέλετε φορέστε ακουστικά λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για τα όσα μας είπατε. Φαίνεται ότι θα είναι μια πάρα πολύ δραστήρια προεδρία δική σας τουλάχιστον από πλευράς Επιτροπής Στεγματικών υποθέσεων έχουμε τόσα θέματα να εξετάσουμε και πολύ σοβαρά με συνέπειες σημαντικότατες του Συμβούλιο. Βασιζόμαστε λοιπόν στις ικανότητές σας να σπρώξετε το Συμβούλιο προσθέσεις. Να προσθέσω ένα ζήτημα που γνωρίζετε καλά. Η Λευκή Βίβλος και πέντε έγγραφα εμβάθυνσης όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης. Οι συζητήσεις από αυτού ίσως δεν θα λήξουν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας, αλλά σίγουρα θα γνωρίζετε τις περισσότερες, θα γίνουν οι περισσότερες εξελίξεις αυτή την περίοδο της Προεδρίας σας. Πώς σκέφτεστε να οργανώσετε τη συζήτηση, όχι μόνο μεταξύ θεσμικών οργάνων, αλλά και μεταξύ Ευρωπαίων ε, πολιτών, μάλιστα από την εμπειρία που έχετε αποκομίσει με την ηλεκτρονική δικυβέρνηση, e-government. Όσον αφορά το θέμα αυτό, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αν θέλετε να συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο διερωτώμε μήπως μπορείτε να προωθήσετε σημαντικά στη συνάντηση στο Ταλίν. Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε το e-citizenship και την e-identity, ηλεκτρονική ταυτότητα και ηλεκτρονική ηθαγένεια των πολιτών. Για να λειτουργήσει όλη η διαδικασία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει κανείς να είναι σίγουρος στην ταυτότητα των ατόμων. Και αυτή η ταυτότητα θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμη σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένα θέμα δικό σας και εμείς περιμένουμε κάτι και ζητούμε κάτι πάνω σε αυτό. Αναφερθήκατε στη διαφάνεια. Εγώ θα έκλεινα επ' αυτού του σημείου τηρώντας το τρίλεπτο που μου διετέθη Σίγουρα πρέπει να έχουμε μια συμφωνία επί της διαφάνειας. Όπως ξέρετε ένα από τα προβλήματα ε, ε, όσον αφορά έχει δισταγμού το Συμβούλιο όσον αφορά αυτό. Δεν αφορά μόνο το ε, μητρό διαφανείας, αλλά όλη τη μέθοδο εργασίας του Συμβουλίου, που είναι πολύ αδιαφάνης. Και σχεδόν κανένας πολίτης ε, στην Ευρώπη δεν ξέρει ότι υπάρχει το Συμβούλιο. Το Συγχέων, το Συμβούλιο με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ε, και είναι άγνωστος ο ρόλος του Συμβουλίου. Διότι τίποτα δεν είναι δημόσιο. Υπάρχει ελάχιστη διαφάνεια. Πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε κάτι σε αυτό το πεδίο. Ευχαριστώ. Ε, thank you. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω Οι συζητήσει για το μέλλον της Ευρώπης ξεκίνησαν τις πιο δύσκολες στιγμές. Πέρυσι. Και ο τρόπος με τον οποίο προχωρήσαμε εμείς ως 27 και στην Πρατισλάβα και στη Ρώμη πραγματικά ήταν πολύ ε, ενδιαφέρον. Τώρα γίνεται μια συζήτηση η οποία τρέχει. Έχουμε τη Λευκή Βίβλο. Έχουμε και τα πέντε έγγραφα προβληματισμού, τα οποία θα έλεγα πως προσφέρουν πάρα πολύ υλικό για προβληματισμό και σκέψη, όχι μόνο σε επίπεδο ακαδημαϊκών και ερευνητικών κέντρων, η think tank, αλλά και σε επίπεδο πολιτικών. Το σχετικό με την παγκοσμιοποίηση, για παράδειγμα, δεν θα έλεγα πως έδωσε επιχειρήματα, αλλά τουλάχιστον ε, χρησιμοποιήθηκε ως ε, τροφή για προβληματισμό για τις συζητήσεις που κάνουμε τον Ιούνιο στο Συμβούλιο και κυρίως για θέματα εμπορικά και για το ποια θα είναι η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμείνει ανοιχτή. Η Προεδρία της Εστονίας θα συζητήσει το έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον της ΟΝΕ στο άτυπο ΕΚΟΦΗΝ που θα γίνει το Σεπτέμβριο και επίσης θα συζητήσουμε και το σχετικό έγγραφο για τον κοινωνικό πυλώνα στην άτυπη συνάντηση του Συμβουλίου Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης τον Οκτώβριο για να δούμε τι θα γίνει με τη μελλοντική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί τρέχουν κάποιες συζητήσεις σε επίπεδο συμβουλίου και αν θέλετε να μιλήσουμε για την ευρύτερη πολιτική συζήτηση είστε και εσείς ερετή πολιτική. και ξέρετε καλύτερα από μένα αυτή τη στιγμή που βρίσκεται η συζήτηση και σε ποιο σημείο είμαστε. Εγώ θα επιμείνω δεν είναι μόνο σημαντικές εδώ οι αλλαγές που θα κάνουμε σε επίπεδο θεσμικών οργάνων. Ίσως ακόμα πιο σημαντικές είναι οι αλλαγές που θα φέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει αυτά τα αποτελέσματα και το μήνυμα αυτών των αποτελεσμάτων να φτάσει μέχρι τους πολίτες. Γιατί αυτό θα κάνει τους πολίτες να αισθάνονται πως η Ένωση είναι πιο σημαντική και ελπίζουμε πως με τον τρόπο αυτό θα ξυπνήσει και το ενδιαφέρον των πολιτών για να συζητήσει κάποια από αυτά τα θέματα. Βεβαίως έχουμε αυτή την ψηφιακή ταυτότητα στην Εστονία ήδη. Ε, έχουμε την ψηφιακή ηθαγένεια και την ψηφιακή ταυτότητα και να σας πω, σας τα προτείνω ένθερμα, γιατί πιστεύω ότι ε, και όλες οι δικλείδες ασφαλείας ε, είναι στη θέση τους και η τεχνολογία υπάρχει και αν θέλετε, εμείς μπορούμε να σας δώσουμε και ε, ψηφιακή άδεια διαμονής, εάν το επιθυμείτε. Αν θεωρείτε δηλαδή ότι θα καταναλώσετε τι αστωνικές ψηφιακέ υπηρεσίε, οπότε υπάρχουν τέτοιου είδου λύσει. Έχουμε την ψηφιακή υπογραφή για παράδειγμα που διευκολύνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την ε, ε, προσωπική αλλά και την επαγγελματική ζωή των ανθρώπων και όπου με τον τρόπο αυτό ε, μειώνει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, μειώνει το χρόνο που χάνει, μειώνει τις προσπάθειες που πρέπει να κάνει, οπότε έχει μεγάλη εξοικονόμηση και υπάρχουν πολλές τέτοιου είδους λύσεις. transparency in various institutions. Uh, Τώρα για τα υπόλοιπα που είπαμε. Υπάρχουν κάποια θεσμικά όργανα που μοιάζουν φοβερά διαφανή, που είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς ε, να καταλάβει τι κάνουν ακριβώς. Στο Συμβουλίο όλοι, όλοι εμπλεκόμενοι, όλοι οι παίκτες εξετάζονται εξονυχιστικά από την κοινή γνώμη στα οικία κράτη-μέλη. Εμείς εκπροσωπούμε τις εθνικές κυβερνήσεις, οπότε η, διαφάνιση, η διαφάνεια, με συγχωρείτε, και το στοιχείο της διαφάνειας είναι πάντα παρόντα. Και γνωρίζουμε σίγουρα για το θέμα της διαφάνειας ποιες είναι οι ανησυχίες. Για το θέμα αυτό έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να προχωρήσουμε και ελπίζουμε πως μέχρι το τέλος της Προεδρίας μας θα έχει δοθεί μια λύση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Πολύ ρεαλιστική η παρουσίασή σας. Τα οικονομικά ζητήματα είναι σημαντικότατα για σας. για τον προστατευτισμό και τους αόρατους φραγμούς για την ελεύθερη αγορά. Πολλοί παρατηρητές σημείωσαν ότι πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν θεσπίσει ανεπίσημους φραγμούς κατά της ενιαίας αγοράς κάποια τέλη όσον αφορά ε, τις μεταφορές, νέα οδηγία για τους εργαζόμενους σε απόσπαση και αυτό επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Η άποψή σας ποια είναι όσον αφορά αυτά τα θέματα. Απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα θέματα που θέσατε είναι ύψης της σημασίας για την λειτουργία της ενώσεώς μας. Η ενία αγορά είναι η καρδιά πολλών τυχών της Ένωσης που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία. Και η ενία αγορά δεν έχει ολοκληρωθεί κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών. Η ενιαία αγορά και ο κοινωνικός πυλώνας είναι αλληλένδετα στοιχεία. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να αναφέρεται κανείς σε κοινωνικά ζητήματα αν ταυτόχρονα γινόταν βήματα για εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και για άρση των διαφόρων φραγμών που εξακολουθούν να εφίστανται όλα τα κοινωνικά ζητήματα στο Συμβούλιο είναι ουσιαστικά προβληματικά, όπως τα περιγράψατε, και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με εξαιρετική προσοχή και με μεγάλη διπλωματία. Και αυτό κάνουμε. Είχαμε πλησιάσει σε επίτευξη ε, θέσεως, κοινής θέσεως του Συμβουλίου για τους αποσπασμένους εργαζομένους δυστυχώς απεδείχθη ανέφικτο τον Ιούνιο. Θα το προωθήσουμε το θέμα. Περίπλοκος τομέας με ελάχιστε αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως και είναι επίμαχο και διχαστικό διότι δεν υπάρχει εξισορρόπηση επιπέδων διαβίωσης και αμοιβών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι δεν πρέπει να υπονομευθεί η ενιαία αγορά. Είναι το κέντρο, η καρδιά πολλών ζητημάτων. Στο Συμβούλιο, στις εργασίες μας, πρέπει να πετυχαίνουμε τη σωστή ισορροπία από πολιτική σκοπιά πόρο απέχει από το να λήξει αυτή η συζήτηση και σας ευχαριστώ που το θέσατε το ζήτημα. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ε, από πλευρά Σάλτε. Θα μιλήσω ισπανικά. Να σας πω πως καταρχήν θέλω να σας καλωσορίσω και να σας πω πως έχουμε στα ισπανικά μία παροιμία που λέει «Από τα ψηλά πέφτουμε στα χαμηλά». Δηλαδή, εντάξει, Ωραία. Κατεβείτε λοιπόν από τα ψηλά να δούμε λίγο τα πρακτικά της καθημερινότητας, γιατί υπάρχουν κάποια θέματα που ανησυχούν ε, εδώ τους ε, ευρωβουλευτές, κυρίως όσους έχουμε ασχοληθεί με τα Panama Papers. Δηλαδή, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ε, πώς μπορούμε να απελευθερώσουμε το δικαίωμα εξέτασης εάν δεν μπορούμε καθόλου να προχωρήσουμε παρόλες προσπάθειες που κάνει ο συνάδελφος Ραμάν Χουαρέκη εκεί. Μας είπατε πως ζούμε σε μία περίοδο όλο αναταράξεις. Ναι, έχετε δίκιο. Δεν μπορούμε εμείς να χορεύουμε μινουέτα και να μην μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί ήταν τεράστιο σκάνδαλο τα Panama Papers και εμάς μας έχετε δέσει τα χέρια και δεν μπορούμε να εξασκήσουμε τις υποχρεώσεις μας εν ώψη των Ευρωπαίων πολιτών και πρέπει να σας πω πως δεν είχαμε τα κατάλληλα εργαλεία για να κάνουμε τη δουλειά μας. Και γι' αυτό θα μας αφήσει το Συμβούλιο να μπούμε στην πράξη και να μην μείνουμε στα λόγια. Και θα επανέλθω σε θέματα της εμπειρίας μας και θα μιλήσω για το Μητρό Διαφάνειας. Θέλω να μας πείτε θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με το Συμβούλιο ή όχι. Γιατί αν δεν μπορείτε, εντάξει, πείτε το, αλλά να το ξέρουμε το συντομότερο δυνατόν, γιατί αυτό που με ανησυχεί είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αποτύχει στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών, αν δεν έχουμε τα εργαλεία να κάνουμε τη δουλειά μας. Και εσείς στο Συμβούλιο δεν μας βοηθήσατε καθόλου. Ευχαριστώ πολύ, ο Υπουργός να απαντήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά το θέμα αυτό για την Επιτροπή για τα έγγραφα του Παναμά, έγιναν ανταλλαγές απόψεων μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Διατείνεστε ότι το Συμβούλιο δεν ήταν συνεργάσιμο. Δηλαδή δεν έδωσε τα έγγραφα που είχε ζητήσει η Επιτροπή. Η θέση του Συμβουλίου ήταν και εξακολουθεί να είναι σας παρακαλώ αποσαφηνίστε το αυτό. Και τα αιτήματα για έγγραφα ήταν πολύ γενικόλογα. Το Συμβούλιο δεν είναι κλειστό όσον αφορά τη συνεργασία μαζί σας για το θέμα οι εκπρόσωποι της Εστονίας θα είναι παρόντες στις ανεπίσημα συνεδριάσεις σας. Είμαστε ανοιχτοί όσον αφορά τη συνεργασία, αλλά πρέπει να επιτευχθεί μια καλύτερη ισορροπία για τη διαφάνεια και το μητρό διαφάνειας. Γνωρίζουμε ότι το βασικό θέμα είναι τι πεδίο καλύπτεται. Τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε. Το Συμβούλιο αποτελείται από 28 κυβερνήσεις και 28 εκπροσώπους κυβερνήσεων. Και πάντα πρέπει να ακολουθήσουν την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές διευθετήσεις για το θέμα αυτό. Η Ιστονική Προεδρία, όπως ανέφερα, έχει στόχο μία λύση. Λύση κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Είμαστε έτοιμοι για συνάντηση πολιτικού επίπεδου το ταχύτερο δυνατόν. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να γίνουν οι δύο πρώτες ερωτήσεις, οι δύο τελευταίες ερωτήσεις μαζί και μετά και οι δύο απαντήσεις. Σας παρακαλώ να είστε σύντομοι. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ καταρχάς για την επίσκεψη που είχατε την ευγένεια να μου επιτρέψετε να κάνουμε στο Στρασβούργο. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ως Επιτροπή ότι ο Υπουργός ενδιαφέρεται για το πόσο έχει προχωρήσει η έκθεση για τις Επιτροπές ε, Έρευνας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Στις 21 Σεπτεμβρίου <coughs> θα συζητήσουν οι τρεις νομικοί σύμβουλοι των τριών θεσμικών οργάνων. Σας παρακαλώ. να προωθηθεί κατόπιν το νομικό κείμενο των τριών νομικών υπηρεσιών, να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση και σας παρακαλώ να ξεκινήσουμε τον ε, τριμερή διάλογο με, με την Επιτροπή και το Συμβούλιο για να δούμε εάν μπορεί να βρεθεί μια λύση για το θέμα αυτό. Επανειλημμένα έχω τονίσει εδώ στην Επιτροπή μας ότι τρία χρόνια τώρα σχεδόν έχει κολλήσει το θέμα, δεν προχωράει. Πέρασαν πέντε προεδρίες που δεν μπόρεσαν να υπερβούν το αδιέξοδο. Και ναι, δεν είναι η ευθύνη αποκλειστικά του Συμβουλίου, αλλά παρόλα αυτά σας παρακαλώ η Εστονία να αποδειχθεί η Προεδρία που δεν ασχολείται μόνο με ψηφιακά θέματα αλλά επιλύει και άλλα. Και όπως είπε και η συνάδελφός μου για να περάσουμε από τις μουσες στο θέατρο. Δεν θέλω μόνο διπλωματική αλλά πολιτική απάντηση. Ως διπλωμάτης, ως διπλωμάτης είστε εξαιρετικός αλλά θέλω να είστε και ως πολιτικά υπεύθυνος. Ευχαριστώ Ραμόν. Η κυρία Τζέιμς και μετά ο Ρίτσο. Δεν λεπτό Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Με συγχωρείτε, δεν ήμουν στην Ολομέλεια την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά διαπίστωσα τι έγινε μετά. Τώρα το λέω βέβαια ίσως ε, ε, ε αλλά θέλουμε να ακούμε τις προεδρίες με τη σειρά τους και να τους δίνουμε σημασία. Αλλά θέλω να αναφερθώ σε θέματα τα οποία κληρονομήσατε από τις προηγούμενες προεδρίες και θα συνεχίσετε να ε, προωθείτε. Αλλά ίσως θα μπορούσατε να περιλάβετε και κάποια άλλα θέματα. Θέματα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους πολίτες, όπως φαίνεται και από τα μέσα. Ποια είναι αυτά να ενταχθούν ταχύτατα ε, οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Τα ελλείμματα του προπολογισμού που θα δημιουργηθούν από τον Brexit. Τι γίνεται με την ε, Ευρωπαϊκή Αμυντική Δύναμη. Και η ενδεχόμενη κατάρρευση της Συμφωνίας Ένωσης Τουρκίας για τον έλεγχο της μετανάστευσης. Αυτό είναι προτεραιότητα για πολλά μέσα. Και τέλος, σας συγχαίρω για αυτά που κάνατε ως εσθονία για τα 5G. Αλλά μήπως μπορείτε να δείτε τι γίνεται και με την ε, κβαντική σύνδεση που επιχειρεί η Κίνα και να επιτύχουν σε διάστημα, σε απόσταση 2.000 μιλίων ε, ασφαλείς ε, επικοινωνίες. Άρα πρέπει και εμείς να καλύψουμε την καθυστέρησή μας. Ο κύριος Κόρμπετ. Λοιπόν, να επανέλθω σε αυτά που είπε ο κύριο Σέπφλιν για τους πολίτες και τον πληθυσμό σε σχέση με τις έδρες. Οι πολίτες της Ένωσης που έχουν πάει σε άλλο κράτος μέλος μπορούν να ψηφίζουν στη χώρα διαμονή τους. Εγώ εκπροσωπώ τους Ούγγρους και Ους που ψήφισαν ε, στο Ιόξια το οποίο εκπροσωπώ. Δεν είναι ότι δεν εκπροσωπούνται, αλλά με προβλημάτισε η ε, πρόσκληση του Υπουργού να γίνουμε όλοι ηλεκτρονικοί πολίτες της Εστονίας. Θα μπορούμε να ψηφίσουμε σε ευρωεκλογές στην Εστονία. Θα μπορούσαμε να είμαστε υποψήφοι. Και αν γίνει το Brexit, θα μπορούσαν πρώην πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν αίτηση για ηλεκτρονική υποψηφιο... Ε, υπηκότητα στην Εστονία και να συμμετέχουν στις εκλογές. Τώρα πιο σοβαρά. Για το θέμα της διοργανικής συμφωνίας. Είπατε ότι το Συμβούλιο κάνει έναν απολογισμό της κατάστασης. Και εμείς το κάνουμε αυτό από την πλευρά μας, ε, με μια ειδική επιτροπή που θα καταλήξει έκθεση. Καλό θα ήταν λοιπόν να συγκρίνουμε πώς έχουμε προχωρήσει, μεν και η Και επίσης, στα πλαίσια της συζήτησης αυτής, αναφερθήκατε στις ε, διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων για την ε, οριοθέτηση, κατεξουσιοδότηση από τις εφαρμοστικές πράξει σα. έδωσαν εντολή συνάδελφοι στο Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Γιατί αυτό είναι το απαραίτητο πρώτο βήμα για να ξεκινήσουν αυτές οι διαπραγματεύσει σοβαρά. Ευχαριστώ Ρίτσον. Λοιπόν, η τελευταία σας παρέμβαση κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ. στον κύριο Χάρη, για την ε, δυνατότητα δημιουργίας εξεταστικών επιτροπών. Έχω την ίδια θέση με εσά. Και εγώ ελπίζω όταν θα ολοκληρωθεί η εργασία των νομικών υπηρεσιών, ελπίζω λοιπόν, να μπορέσουμε να εξετάσουμε εάν και κατά πόσον υπάρχει περιθώριο συμφωνίας. Αυτό άκουσα ότι είπατε. Και αυτή είναι σωστή περιγραφή της φάσης στην οποία ευρισκόμαστε. Προς την κυρία Τζέιμς. Πολύ σωστά τα θέματα που αναφέρατε και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωσή μας σε αυτή τη συγκυρία. δεν τις ανέφερα στις αγωγικές μου παρατηρήσεις γιατί εστίασα περισσότερο στα θέματα που είναι κυρίως αρμοδιότητες της Επιτροπής σας, της ΑΦΚΟ. Όλα τα θέματα που αναφέρατε είναι από τις προτεραιότητες της ε, Εστονικής Προεδρίας. Αλλά κάτι για την κυβερνοάμυνα η Εστονία ήταν η πρώτη κυβέρνηση που υπέστη στοχευμένη επίθεση το 2007. Άρα εξαγάμε κάποια διδάγματα στον τομέα αυτό. Στις πρόσφατες ε, κύβερνο επιθέσεις παγκοσμίως η Εστονία Εφήγη σχετικά λίγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Σεπτέμβριο με μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια που θεωρούμε ότι θα είναι αναλυτική και ότι θα περιέχει συγκεκριμένες ενέργειες. Η Εστονική Προεδρία βεβαίως κατόπιν θα κινηθεί σύντομα και θέλουμε να εγκρίνουμε συμπεράσματα το Νοέμβριο για το θέμα αυτό. Κύριε Κόμπετ, ε, λυπάμαι, αλλά θα σας απογοητεύσω. Η ηλεκτρονική άδεια διαμονής δεν σας δίνει δικαίωμα ψήφου. Μπορείτε να ψηφίσετε στις ευρωεκλογές και στις τοπικές εκλογές στην Εστονία ως πολίτης τρίτης χώρας αλλά πρέπει να έχει ζήσει κανείς στην Εστονία για συγκεκριμένο χρόνο, χρονικό διάστημα, κάποια χρόνια. αλλά μπορείτε να αξιοποιήσετε διάφορες ψηφιακές υπηρεσίες. για τις κατεξοδότηση και εφαρμοστικές πράξεις. Βεβαίως είμαστε διαθέσιμοι να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να εξετάσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι αυτό που διαπιστώνουμε και εμείς είναι αυτό το οποίο είναι πως έχετε τη δυνατότητα να δείτε και την ευρύτερη εικόνα και μπορείτε και να ε, παραδώσετε τα απαραίτητα, οπότε αυτό είναι πολύ αισιόδοξο εν ώψη της Προεδρίας σας. Για όσους μας ζητάνε ε, να προσφέρουμε και να συνεισφέρουμε στη συζήτηση το κάνουμε. Αν έχετε οποιαδήποτε επιθυμία, ε, παρακαλώ πολύ ε, να αισθανθείτε ελεύθερα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ε, το κομμάτι της συνεδρίας με τον Υπουργό έχει τελειώσει. Θα μείνουμε εμείς εδώ για τις ψηφοφορίες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι κυρία Πρόεδρε και τους συναδέλφους για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με στοχευμένες και καλά τεκμηριωμένες ερωτήσεις. Η Προεδρία είναι στη διάθεσή σας.

Dear colleagues, can, I, can we immediately move to the next point? Να πάμε αμέσως στο επόμενο σημείο που είναι οι ψηφοφορίες, αγαπητοί συνάδελφοι. And also, so you're waiting. I think there is another one. I'm told we still see people who I don't know where you keep those cards that you don't have them with. Δεν καταλαβαίνω πού βάζετε τις κάρτες σας και τις ξεχνάτε, λέει η πρόεδρος. κύριο Μέτρη, δεν έχει την κάρτα του, κάποιο άλλο μπορεί στον κάτω-κάτω να μην τη χρειαστούμε. Άλλο κανεί έχει μείνει χωρί κάρτα. Σα παρακαλώ να μα ενημερώσετε. Για παρακαλώ να μετρηθούμε, να ελέγξουμε το σύστημα. Παρακαλώ να τοποθετήσετε τι κάρτε στο μηχάνημα. Ξεκινάμε. Uh, we are making... We are checking the ελέγχουμε τα μηχανήματα, ελέγχουμε ότι έχετε τις κάρτες Σα Σας παρακαλώ πολύ χρησιμοποιήστε τα μηχανήματα για να κάνουμε τον έλεγχο. In this um, oh, Okay, two, two colleagues put their cards but they don't vote, so I assume we assume that uh, every... Δύο συνάδελφοι δεν έχουν ε, βάλει κάρτα στο μηχάνημα. 22, 22 είμαστε. Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν. Μιλάμε για το σχέδιο για το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οικονομικό έτος 2018. Να ξεκινήσουμε. Τροπολογία πρώτη, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1,1, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2,1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 τι είναι αυτό Λοιπόν, τώρα είναι τα πειρωματικά σχέδια, άρα λοιπόν ελεύθερη ψηφοφορία, δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα υπέρ. Στην 5 κατά αποχές εγκρίνεται, 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 4,1 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ Υπέρ για την 9. Ψηφίζουμε την 9. Υπέρ. Κατά. Μπορούμε ηλεκτρονικά παρακαλώ πολύ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Λοιπόν, 17-6 εγκρίνεται. Δεν σας ακούω. Ό,τι και να πείτε δεν άκουσα. Θέλετε, έχετε αντίρρηση για το αποτέλεσμα, φωνάξτε το. 3,1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5,1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ με την προφορική τροπολογία που δεν θα βάλουμε substantial, θα βάλουμε το όχι ουσιαστικό αλλά κατάλληλο. Ωραία. Λοιπόν, όπως τροποποιήθηκε για την 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Φτάνουμε λοιπόν στην τελική ψηφοφορία για το σχέδιο. Θα το κάνουμε ονομαστικά. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. 19-4. Εγκρίνεται λοιπόν. Ξέρετε κι εσείς το 12 δεν θα το ψηφίσουμε. Ζήτησε ο Πασκάλ Ντιράν ε, περισσότερο χρόνο για τις τροπολογίες. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο σημείο 13 που είναι το ψήφισμα, συγγνώμη, ο κανονισμός για το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Κανονισμό 1141, κάθετος 2014, καθεστώ και χρηματοδότηση ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων. Εδώ έχουμε την ανταλλαγή απόψεων για την ενδεχόμενη αναθεώρηση αυτού του κανονισμού. Έχουμε καλέσει για αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών τον Ράινερ Βιλάντερ, που είναι υπεύθυνο για τα πολιτικά κόμματα, αντιπρόεδρος όπως επίσης τον κύριο Κλετή που είναι από την DG Finance από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον κύριο Γιώχανσον που είναι αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Μίκαελ Άνταμ από ε, το από την αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ιδρύματα και θα μιλήσουμε για τα θέματα αυτά, θα ακούσουμε τις απόψεις σας, τι γίνεται με τα πολιτικά κόμματα και τα ιδρύματα. Ξέρετε και εσείς πως είναι μεγάλη η ιστορία αυτής της υπόθεσης και έχουμε οδηγηθεί σε μια συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα και θα μιλήσουμε παράλληλα και για την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Κοινοβουλίου. Έχουμε υποβάλει και μια προφορική ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου έχουμε όλα τα αιτήματα ε, και τα ερωτήματα που, στα οποία έχουμε καταλήξει. Το ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 15 Ιουνίου μετά τη συζήτηση. Οπότε θα ήθελα τώρα να καλέσω τους ομιλητές. Θα ήθελα να ξεκινήσω καταρχήν με τους δύο αντιπροέδρους. Βέβαια βλέπω μόνο έναν, ελπίζω πως θα είμαστε δύο. Δεν βλέπω την κυρία Λούνατσεκ. Ωραία, Ράινερ. Παρακαλώ πολύ, θα ήθελα ο κύριος Ράινερ Βίλαν να ξεκινήσει τη συζήτηση με την παρουσίαση που έχει να μας κάνει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε και σε επίπεδο επιτροπή Έχουμε συζητήσει επιτροπή, έχουμε ψήφισμα του Κοινοβουλίου, έχουμε ανταλλαγή ε, επιστολών μεταξύ των κομμάτων που θεωρούν όλοι ότι πρέπει να υπάρξει ταχεία βελτίωση. Στην αρχική έκθεση Γιαννάκου ε, προβλεπόταν το 2018 αυτή η βελτίωση αλλά θεωρώ ότι ε, αν αρχίσουμε να συζητάμε και να ψηφίσουμε το θέμα αυτό το Γενάρη του 2018, τότε μέχρι τον ε, Οκτώβριο δεν θα έχουμε τελειώσει. Οπότε θα χάσουμε και τον επόμενο χρόνο, γιατί αρχές του επόμενου χρόνου πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες προκηρύξεις για να αλλάξει η κατάσταση. Οπότε πρέπει να, να εργαστούμε πολύ ε, εντατικά για το κείμενο αυτό της Κομισιόν. Ε, το είχαν ανακοινώσει πριν τις διακοπές, ελπίζω να το υποβάλουν αμέσως μετά τις διακοπές και ελπίζω να τα αντιμετωπίσουμε αυτά ούτως ώστε να έχουν εγκριθεί και να μπορούν να εφαρμοστούν οι νέοι κανόνες για τις εκλογές του 19. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποφύγουμε την προσπάθεια να γίνει ουσιώδης βελτίωση. Αν ξεκινήσουμε αυτή την αποτίμηση ήδη πριν τώρα το 18, θα πρέπει να κάνουμε τα απολύτως απαραίτητα βεβαίως, αλλά κατόπιν θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ήδη από το φθινόπωρο του 19 ή το νωρίτερο, αρχές του 20, θα πρέπει να γίνει μια θεμελιώδης συζήτηση για αυτούς τους κανόνες και θα έχουμε ήδη τότε και τα πρώτα αποτελέσματα από τη λειτουργία τους. Θεωρώ ότι πρέπει λοιπόν να βελτιωθούν εκ βάθρων τα πράγματα. Αλλά αν το επιχειρήσουμε τώρα δεν θα προλάβουμε, γιατί μας πιέζει πολύ ο χρόνος. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα τα εξής τρία θέματα, όπου έχουν υπάρξει προβλήματα ήδη. Πρώτα απ' όλα, δεν θα, είναι, δεν θα πρέπει στο μέλλον να είναι δυνατό να είναι κανείς μέλος πολλών κομμάτων. Αυτό ήταν κάτι που δεν προβλέψαμε. Ιδίως από βουλευτές οι οποίοι εξελέγησαν με ένα ψηφοδέλτιο που δεν ανήκε σε καμία πολιτική οικογένεια και υπάρχουν σαφείς κανόνες. Και είδαμε ότι υπάρχει ε, περιθώριο για καταχρήσεις. Το δεύτερο, ότι τα κόμματα θα πρέπει να έχουν ευρωπαϊκή διάσταση και γι' αυτό θα πρέπει λοιπόν να αυξηθεί το ελάχιστο όριο για τη δημιουργία τους, που τώρα είναι ένας μόνο βουλευτής ανακόμα. Αυτό θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης, θα πρέπει να μειωθεί η υποχρέωση συγχρηματοδότηση από 15% στο 7,5%. Και να εφαρμοστεί αυτή η τροποποίηση. Αυτές είναι λοιπόν οι προτάσεις μου. Πρέπει να εφαρμοστούν τάχιστα το Προεδρείο μέχρι του χρόνου τον Απρίλιο πρέπει να έχει κάνει τις αναγκαίες προκηρύξεις με νέα βάση εν ώψη του 19. Και όσο πιο γρήγορα γίνεται να γίνουν τα επόμενα βήματα θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εφαρμοστούν όλα αυτά πριν το φθινόπωρο του 18 εάν περιορίσουμε την αντιπαράθεση για να μπορέσουμε να τα εφαρμόσουμε στην επόμενη θητεία να έχουμε επαρκή χρόνο, να έχουμε συλλέξει εμπειρίες οι οποίες θα μας επιτρέψουν να περάσουμε στα περαιτέρω βήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Ράινερ. Η Ουλρίκη κατέφθασε εγκαίρως. Ελπίζω να έχει ανακτήσει την ανάσα της και να πάρει το λόγο. Θα δώσω το λόγο στο δεύτερο αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, την κυρία Ουλρίκη Λούνατσεκ. Έχετε το λόγο. Συγγνώμη, ναι, που καθυστέρησα. Καταρχάς, Ευχαριστώ την Επιτροπή ΑΦΚΟ που οργάνωσε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι παρούσα και συνεργάζεται μαζί μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Με τον συνάδελφό μου, τον Ράινερ Βίλαντ, έχουμε εξεργαστεί το θέμα για κάποιο χρονικό διάστημα και όπως εξήγησε πρέπει να προσέξουμε κάποια σημεία ώστε το όλο ζήτημα να προωθηθεί καλύτερα από ό,τι πριν. Υπάρχουν κάποια κενά που πρέπει να καλυφθούν, που ανακαλύψαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Και κατά την άποψή μου υπάρχουν τρία πράγματα τα οποία θα ήθελα να τονίσω σε αυτή τη σύντομη παρουσίαση. Πρώτα απ' όλα ανακαλύψαμε εδώ και δύο-τρία χρόνια ότι ένα από τα κενά ήταν το εξή. Εάν ένα κόμμα σε ένα κράτος μέλος δεν είναι μέλος Ευρωπαϊκού Κόμματος τότε οι βουλευτές του μπορούν να υποστηρίξουν διαφορετικά. Οι ευρωβουλευτές του μπορούν να υποστηρίξουν διαφορετικά πολιτικά κόμματα. Και μπόρεσαν δύο ευρωπαϊκά κόμματα να φτάσουν στο όριο για να πάρουν το όριο για δύο, παρόλο που έχουν εκλεγεί από, από ένα κόμμα. Κοιτάξτε, εμεί δεν είχαμε σκεφτεί ότι κάποιο θα το κάνει αυτό. Συνέβη. Είναι ένα κενό το οποίο πρέπει να καλυφθεί. Κάτι άλλο. Και είναι σημαντικό να εξετάσουμε το όριο. Πόσοι βουλευτές χρειάζονται για να σχηματιστεί ένα κόμμα. Υπάρχουν διάφοροι αριθμοί που κυκλοφορούν. Εγώ θα έλεγα ότι θα σας παρακαλούσα να λάβετε υπόψη ότι έχουμε υπάρχουν κάποιοι από μικρότερη πολιτική ομάδα, μικρότερο κόμμα όπως εγώ, είναι σημαντικό να μην είναι υψηλό Ένα, δύο. Για μένα ε, αυτό είναι το κατάλληλο επίπεδο. Βέβαια υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις. Για να εξασφαλίσουμε όμως ότι πραγματικά υπάρχει ευρωπαϊκό πνεύμα, ευρωπαϊκός χαρακτήρας, κάτι που αναφέρατε σε κύριε Βίλαντ, αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να επικρατεί διαφάνεια σχετικά με το ποια είναι τα εκλεγμένα μέλη σε διάφορα επίπεδα για τα ευρωπαϊκά κόμματα. Όχι μόνο εκείνοι που καθιστούν επιλέξιμο αυτό το κόμμα για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αλλά και εκείνους που εκλέγονται και στηρίζονται σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο. Ε, διότι μέχρι τώρα αυτό δεν έπαιζε ρόλο. Ο κάθε άνθρωπος που εκλέγεται σε οποιοδήποτε επίπεδο είναι μια δημόσια προσωπικότητα ε, και θα πρέπει να γνωστοποιεί το όνομά του ή το όνομά της. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι, δεν θα πρέπει να είναι άγνωστοι. Το συζητήσαμε και πριν. Αυτός εξευρωπαϊσμός των ευρωπαϊκών κομμάτων πρέπει να φροντίσουμε ότι εκείνοι που υποστηρίζουν τα ευρωπαϊκά κόμματα ή τα ιδρύματα θα πρέπει να εφαρμόζουν τη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων, να την υποστηρίζουν, να είναι μαζί μας, στο πλευρό μας, να εστερνίζονται τα όσα εκπροσωπεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα πρώτα μου εισαγωγικά σχόλια και προσβλέπω σε μια καλή συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ Ουλρίκε. Ο κύριος έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε που είμαι επιφερτασμένος για τα χρήματα που, τις φορές που καταβάλλονται στα ιδρύματα να παρουσιάσω κάποια επιχειρήματα όσον αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού του 2014. Αυτές οι πληροφορίες που θέλω να σας δώσω επικεντρώνονται επί των προτεραιοτήτων της αναθεωρήσεως και της επιθυμίας βελτίωσης. Αυτό που ανέφεραν ε, οι δύο ε, αντιπρόεδροι. Αλλά θα ήθελα να παρουσιάσω την άποψη της Γενικής Διεύθυνσης των Οικονομικών όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τον ετήσιο έλεγχο των λογαριασμών των πολιτικών κομμάτων και των ε, ιδρυμάτων των ευρωπαϊκών. Λοιπόν, συμφωνώ με τα τρία σημεία που είχαν προτεραιότητα, ίσως κάπως διαφορετική σειρά θα παρουσίαζα εγώ. Θα ήθελα να προσθέσω δύο άλλα στοιχεία τα οποία είναι κάπως δευτερευούς σημασίας αλλά που πρέπει να λάβουμε υπόψη στην αναθεώρηση. Οι αντιπρόεδροι αναφέρθηκαν στη δυσκολία των κόμματων να έχουν επαρκείς ιδίους πόρους και κάποια να κάποιες παρατυπίες που διαπιστώθηκαν στον αφορά τη χρηματοδότηση και να υπάρχουν επαρκείς ίδιοι πόροι. Ο είναι ότι ένα κόμμα θα πρέπει να έχει 15% ιδίους πόρους και ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως συμβάλλει το 85% όσον αφορά τις ε, νόμιμες δαπάνες που ε, πραγματοποιούνται. Όλα τα κόμματα έχουν λίγο πολύ δυσκολία να έχουν επαρκείς εισφορές, να τις συλλέξουν, να τις πράξουν στο βαθμό που έχει εντατικοποιηθεί η προσπάθεια των, ε, τα τελευταία 10 χρόνια στον προπολογισμό. Τα, τα εθνικά κόμματα έχουν φτάσει στα όρια της χρηματοδότησης που μπορούν ε, να έχουν ή τα εισφορές που δίνουν τα μέλη στα κόμματά τους, ενώ τους απαγορεύεται από την άλλη πλευρά να χρηματοδοτηθούν από άλλες οδούς, διότι οι δωρές είναι στα 12.000 ευρώ μέχρι 18.000 ευρώ ε, στο νέο καθεστώς, 12 στο παλιό, 12.000. Λοιπόν, είτε κάποια κόμματα κάνουν κάποιους ελιγμούς δανειοληπτικούς και ο εξωτερικός ελεγκτής κάθε χρόνο μας παρουσιάζει στο, στον, ε, τις δραστηριότητες, τις συνεχιζόμενες συναλλαγές. Εάν έχουν δοθεί κάποια καινούρια χρήματα σε αυτά τα κόμματα, θεωρείται ε, ότι έχουν χροκοπήσει λόγω της μεγάλης ευαισθητοποίησης που δείχνουν στον φάτη χρηματοδότηση ή αν έχουν σωρεύσει χρέη από τη διανοληψία. Δεύτερο πρόβλημα είναι η κατάχρηση ε, με μια συνεισφορά διαφορετικού είδους ε, που είναι δύσκολο να ελεγχθούν και τα διάφορα κείμενα είναι δύσκολο να γίνουν σεβαστά διότι οποιοδήποτε μπορεί σε είδους να δώσει συνεισφορά και η αξιολόγηση αυτών των συνεισφορών είναι δύσκολο να αποτιμηθεί, δύσκολο να ελεγχθούν. Τέλος ανακαλύψαμε και κάποιες πρακτικές πολύ αμφισβητήσιμες, διότι υπάρχουν συγκρούσεις προφανής συμφερόντων ε, μέσω μια επιχείρηση Φερρυπίν ε, 10-15 του πληρώνει κάποια χρήματα και 10-15% από ένα, από ένα διαγωνισμό που κερδίζει μια εταιρεία ε, καταβάλλεται. Λοιπόν, αυτό μας οδήγησε και μας οδήγησε την ΟΛΑΦ να διαπιστώνει ε, ότι υπάρχουν τέτοια προβλήματα συγκρού συμφερόντων και έχει προσφύγει στο δικαστήριο. Ποια είναι η λύση που μπορούμε να βρούμε. Η Αντιπρόεδρος έκανε μια πρόταση 7,5% μια μείωση, 5% οι ίδιοι πόροι. Η ιδέα είναι να υπάρξει δημόσια χρηματοδότηση, ανοιχτή χρηματοδότηση αυτών των κομμάτων να ε, επιβάλλουμε μια ε, χρηματοδότηση από ιδίως πόρους που είναι δύσκολο να επιτευχθεί, ίσως είναι ένας περιορισμός διότι στο χρηματοδοτικό κανονισμό έχουμε την αρχή της χρηματοδότησης αλλά πρέπει να γίνει παραλυσμός με τη δημόσια ανοιχτή χρηματοδότηση. Μετά η χρηματοδότηση των πολύ μικρών κομμάτων ή πολιτικής, κάποιες πολιτικής λέσχης. Βλέποντας από κοντά αυτό το θέμα, δύσκολο να πετύχουν τους στόχους που έχουμε θέσει, δηλαδή να ε, συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά την ευρωπαϊκή ε, συνείδηση. Αν υπάρχει ένας βουλευτής, 7 μέλη ενός Εθνικού Κοινοβουλίου, Περιφερειακού Κοινοβουλίου και εν συνεχεία οι πόροι που συλλέγονται απλώς κατανέμονται για πολιτικές δράσεις των μελών. Δύσκολο είναι να μιλήσει κανείς ότι αυτό αποτελεί Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα, Ευρωπαϊκό ε, Ίδρυμα. Έχουμε έξι κόμματα που έχουν λιγότερους από ευρω... Ε, πέντε ευρωβουλευτές. Όπως έλεγε η Αντιπρόεδρος η κυρία Λούνατσεκ, το θέμα είναι να δούμε κατά πόσο μπορούμε να αυξήσουμε, αν πάμε στους τρει όσον τον ελάχιστο αριθμό, αυτό δεν αλλάζει τίποτα, τον αριθμό των μέλων. Αν το ελάχιστο ήταν 7 μέλη, θα είχαμε 5 κόμματα μικρού μεγέθους που θα εξαφανιζόταν και αν εφηγραμμιστούμε με τον κανόνα των πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου, δηλαδή 25, θα είχαμε και άλλες συνέπειες. Υπάρχει μια άλλη λύση για να αποφύγουμε αυτό το το πρόβλημα της χρηματοδοτήσεως των πολύ μικρών κομμάτων, αυτό που η κυρία Λούνατσεκ ε, ανέφερε προηγουμένως. Να μειώσουμε το σταθερό κομμάτι που δίνουμε, το πάγιο κομμάτι που δίνουμε σε κάθε κόμμα, 32 εκατομμύριο διαθέσιμα χρήματα πηγαίνουν κατά 15% σε κάθε κόμμα και συνεχεία αναλογικά με τους ευρω... ευρωβουλευτές. Αυτό σημαίνει ότι με 15-16 κόμματα κάθε κόμμα το οποίο ε, παρουσιάζεται μπορεί να πάρει 300.000 ευρώ σαν βάση για 40.000 ευρώ αναβουλευτή που προστίθεται. Αυτή η περίπτωση που ανέφερε η κυρία Λούνατσεκ. Δύο βουλευτές του ίδιου Εθνικού Κόμματος που πηγαίνουν σε δύο ευρωπαϊκά κόμματα, αν προσθέσουμε και τα ευρωπαϊκά ιδρύματα, μπορεί να έχει κανείς δύο φορές τη βάση και δύο φορές 40.000 ευρώ αναλογικά να βουλευτεί. Αν μειώναμε λοιπόν 15% και το πηγαίνουμε στο 5-0% και αν κάναμε μια κατανομή αναλογική όπως γίνεται για τις πολιτικές ομάδες εντός του Ευρωκοινοβουλίου θα έλεγα το κίνητρο για τη δημιουργία κόμματος για 40.000 ευρώ ε, θα ήταν πολύ μικρότερο και τρίτη λύση θα ήταν να περιορίσουμε τα ευρωπαϊκά κόμματα και έρχομαι εδώ στο τρίτο πρόβλημα που ανέφερε ο κύριος Βίλαντ, ο, όσον αφορά τις διασυνδέσεις, παράλληλες συμμετοχές. Στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει να συμμετέχουν μόνο εθνικά κόμματα, όχι μέλη απομονωμένα. Α, αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να αξιολογηθεί και θα πρέπει να υπάρξουν ευρωπαϊκά κόμματα που να αποτελούν το άθροισμα των εθνικών κομμάτων μελών που δε, μετράνε όμως και ανεξάρτητους πολίτες αμήλυτους. Αυτό θα ήταν εποφελές και για το τέταρτο σημείο που θέλω να αναφέρω. Όσον αφορά τις ευθύνες, τις βασικές ποινικέ του αστικού κώδικα, τις ευθύνες που απορρέουν για αυτά τα κόμματα. Έχουμε τρία κόμματα και τρία ιδρύματα ε, που ε, έχουν χρεοκοπήσει και έχουν μπει σε ρευστοποίηση διότι έπρεπε να επιστρέψουν κάποια ποσά στο Ευρωκοινοβούλιο διότι δεν ήταν νόμιμες οι δαπάνες. Αυτό το πρόβλημα αυξήθηκε με τη νέα νομοθεσία, με τον νέο κανονισμό που θα έχουμε προχρηματοδότηση 100%. Δεν θα παραμένει κανένα απόθεμα μετά την ε, εξέταση των λογιστικών στοιχείων είναι νομική δομή που οικοδομείται επί ε, μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί η ευθύνη του Προέδρου, του υπεύθυνου για τα, του Ταμεία κλπ. Ε, αλλά το όλο μονοπάτι είναι μακρύ. Αν υπήρχαν ευρωπαϊκά κόμματα που αποτελούνται μόνο από εθνικά κόμματα, εκεί θα, έλεγα, θα είχαμε ε, μία πηγή προσφυγών σε περίπτωση μη χρηστής διαχείρισης ή απατών. Θα ολοκληρώσω ε, με δύο άλλα σημεία. Τα ευρωπαϊκά κόμματα, ε, κάποιοι γενικοί γραμματείς αυτών είναι εδώ, έχουν πρόβλημα να βρουν κονδύλια για τη χρηματοδότηση εκστατιών για δημοψηφίσματα που απαγορεύονται αλλά ε, εξεφράστηκε κάποια επιθυμία να μπορούν αυτό να το κάνουν όταν πρόκειται περί ευρωπαϊκών ζητημάτων που τίθενται σε δημοψήφισμα. Και τέλος ο κύριος Βίλεντ αναφέρθηκε σε ε, reporting που θα πρέπει να γίνει στα μέσα του 2018. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να εξακολουθήσουν να επανεξετάζονται και να γίνουν κατάλληλες προτάσεις. Εάν η αναθεώρηση που εξετάζεται υλοποιηθεί, μόλις το 2019 θα δώσει αποτελέσματα και το πραγματικό τελικό αποτέλεσμα κλείσιμο θα λάβει χώρα το 2020 και πραγματική έκθεση για τα νέα μέτρα τα οποία τώρα συζητούμε δεν θα είναι χρήσιμο να γίνει παρά μόνο τις αρχές του 2021. Αυτό βέβαια δεν μειώνει σε τίποτα την ανάγκη να ξεκινήσει ένας προβληματισμός στα μέσα του 2018 για όλα τα άλλα ζητήματα τα οποία δεν ε, έχουν εξεταστεί εδώ φέστο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω ε, την κυρία Γιώχενσεν αν θέλει να πάρει το λόγο. Ξέρω πως ε, σας έχουμε δει και στο παρελθόν. Κυρία Γιώχανσεν, σας παρακαλώ πολύ να σας πω πως είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Ε, θα ήθελα να σας πω ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς στηρίζουμε πάρα πολύ αυτή την προσπάθεια που γίνεται και συμμετέχουμε στο, στη συζήτηση αυτή για τα πολιτικά κόμματα και τα ιδρύματα στην Ευρώπη και όλα τα σχετικά ζητήματα. Εμείς παρακολουθήσαμε και καταγράψαμε όλα τα θέματα τα οποία προέκυψαν από τη συζήτηση το Μάρτιο, όπως επίσης και στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Και εμείς έχουμε δείξει πως είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μια διαδικασία με το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να διαπιστώσουμε πώς λειτουργούν στην πράξη οι νέοι κανόνες. Να σας υπενθυμίσω τον κανονισμό του 2014 που έχουμε σημαντικές ε, καινοτομίες, ε, που έχουμε θέσει δικλείδες ασφαλείας και που θέλουμε με τον τρόπο αυτό να γίνουν σεβαστές οι βασικές ε, ευρωπαϊκές αρχές από όλους όσους έχουν καταγραφεί και να σας πω πως η πρόσφατη εμπειρία που έχουμε από τη λειτουργία του τρέχοντος συστήματος μας έχει δώσει την ε, δυνατότητα και ιδέες για να προτείνουμε μία ε, νέα ε, εκλέπτυνση του συστήματος πριν τις εκλογές του 19 και μάλιστα έχουμε βεβαιώσει πως επιθυμούμε προς αυτή την κατεύθυνση να εργαστούμε παρόλο που όλοι γνωρίζουμε ότι αυτός είναι ένας φιλόδοξος στόχος Και θα πρέπει οι αλλαγές αυτές να είναι στοχευμένες, να συνεργαστούμε έτσι ώστε να προετοιμάσουμε το πολιτικό έδαφος και να έχουμε επαρκή στήριξη όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου αλλά και στο Συμβούλιο. Είμαστε λοιπόν σίγουρα δεσμευμένοι προς αυτή την κατεύθυνση και οι συζητήσεις σήμερα θα παίξουν και αυτές το ρόλο τους. Θα είναι ε, μια ε, συνεισφορά χρήσιμη στα όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των προτάσεων που καταθέτει και πρέπει να σας πω πως σήμερα ο ρόλος μου είναι κυρίως να σας ακούσω. Να ακούσω προτάσεις, να ακούσω σχόλια και δεν μπορώ βέβαια να προδικάσω ποια θα είναι η τελική απόφαση που θα λάβουν οι επίτροποι. Αυτό όμως που μπορώ να σας εξασφαλίσω είναι πως εμείς είμαστε σαφέστατα δεσμευμένοι ε, και θα εξετάσουμε όλα τα σημεία που ανέφεραν οι ε, αντιπρόεδρε, η συγχρηματοδότηση, ελάχιστο κατόφλι, οι ε, πολιτικά κόμματα και όλα όσα ανέφερε και ο Γενικός Διευθυντής. Οπότε, το μόνο που μπορώ να πω κλείνοντας είναι πως εμείς, εμείς στηριζόμαστε σε όσα λέει, κάνατε εσείς για να δημιουργήσουμε και αυτό το ε, σφριγιλό πολιτικό περιβάλλον στην Ευρώπη που όλοι επιθυμούμε και με χαρά θα ακούσω τη συζήτηση σήμερα. Θα ήθελα να ζητήσω τώρα τον ε, Διευθυντή της Αρχής για τα Ευρωπαϊκά Κόμματα και τα Ιδρύματα να μας κάνει την παρουσίασή του. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που με καλέσατε και μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω και τις ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην πράξη με το καινούργιο σύστημα για εμείς στην αρχή και φαντάζομαι πως πρέπει να ξεκινήσω λέγοντας πως η αρχή αυτή είναι σχετικά καινούρια. Μας ε, ε, δημιούργησαν πέρσι το Σεπτέμβριο. Είναι μάλλον περιορισμένα τα στοιχεία τα οποία έχουμε συλλέξει για να μπορούμε να αξιολογήσουμε τις πρακτικές επιπτώσεις της δράσης μας. Παρ' όλα αυτά, με τις εφαρμοστικές διαδικασίες έχουμε αποκτήσει κάποια εμπειρία, την οποία θα προσπαθήσουμε να μοιραστούμε μαζί σας σήμερα. Θα ξεκινήσω με μια γρήγορη αναδρομή στο καινούριο σύστημα και τον κανονισμό. Είχα σκοπό να μιλήσω για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της αρχής, αλλά επειδή οι προλαλήσαντες ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένοι, εγώ αυτές τις διαφάνειες θα τις περάσω στα γρήγορα, θα κοιτάξω το κομμάτι που αφορά το που βρισκόμαστε σήμερα και μετά θα κάνω και κάποιες παρατηρήσεις για ενδεχόμενη νομική αναθεώρηση, λαμβάνοντας υπόψη τα πρακτικά ζητήματα που αποσχολούν την αρχή μας. Ξέρετε κι εσείς πως ο νέος κανονισμός εφαρμόστηκε από 1η Ιανουαρίου τρέχοντος και δημιούργησε μια νέα αρχή την οποία εκπροσωπώ εγώ εδώ σήμερα. Είναι ανεξάρτητα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συστήθηκε έτσι ώστε να κατοχωρηθούν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα και να επαληθεύσει το κατά πόσο συμμορφώνονται με τους τρέχοντες κανόνες και να επιβάλλει κυρώσεις σε περίπτωση που δεν έχει ε, συμμορφωθεί κάποιος. Έχουμε λοιπόν έναν διοικητικό υπάλληλο, έναν νομικό και θα περάσω μετά τις επόμενες δύο διαφάνειες κάνοντας μόνο μία παρέμβαση, τα όσα είπε η κυρία Λούνατσεκ προηγουμένως για τη διαφάνεια, να σας πω πως για τη διαφάνεια ο νέος κανονισμός αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Στο διαδίκτυο εμείς θα βάλουμε όλες τις αιτήσει που μας υποβάλλονται με τους φακέλους που τη συνοδεύουν και νομίζω ότι αυτό αποτελεί μεγάλη πρόοδο σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα. Έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια σήμερα, όχι ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, αλλά νομίζω ότι το καλό θετικό στοιχείο του νέου συστήματος ε, είναι ακριβώς αυτό και διαφέρει από το προηγούμενο. Για το πού έχει η κατάσταση. Να σας πω ότι ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο και έχουμε συμφωνήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώ θα κατανείμουμε τι εργασίε μα γιατί η δική μα ε, προσπάθεια είναι συμπληρωματική στο όσο έχει κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. διαδικασία καταχώρηση ξεκινήσαμε από τον Ιανουάριο προετοιμάζοντα τη διαδικασία με κατευθυντήριε γραμμέ προ του ετούντε και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη μέση τη διαδικασία και κοιτάμε ένα καλό νούμερο αιτήσεων και από το Σεπτέμβριο και μετά θα κάνουμε μια ενημερωμένη εξέταση του θέματος της χρηματοδότησης, έτσι ώστε να γνωρίζει το Κοινοβούλιο τι χρηματοδότηση χρειάζεται και να ε, θα στείλουμε τις προφορίες αυτές στο Κοινοβούλιο και από του χρόνου θα κοιτάμε να υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με όλους τους χρηματοδοτικούς κανόνες που είναι στον κανονισμό. Έτσι λοιπόν θα προστατεύσουμε και εμείς και θα συνεισφέρουμε στο σύστημα. Έχουμε λάβει τρεις αποφάσεις, έχουμε καταχωρήσει τρία ευρωπαϊκά κόμματα τους φιλελεύθερους, το ΕΛΚ και τους σοσιαλιστές. Έτσι λάβαμε τις, με αυτή τη σειρά λάβαμε τις αιτήσει. Έχουμε άλλα έξι κόμματα που είναι, έχουν υποβάλει επίσημη αίτηση και είναι σε κρεμότητα. Και δύο ε, εκκρεμεί αιτήματα από ιδρύματα. 15 ε, περίπου σχέδια αιτήσεων έχουν ε, κατατεθεί. Εμείς ξεκινήσαμε μια άτυπη διαδικασία για να διευκολύνουμε όσους θέλουν να αιτηθούν, έτσι ώστε να γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, αλλά οι επίσημες αιτήσεις που λάβαμε με αυτές τις οποίες ανέφερα προηγουμένως. Και βέβαια τα χρονοδιαγράμματα είναι αρκετά σφιχτά. Και νομίζω ότι η αλλαγή του συστήματος αποτέλεσε πρόκληση για όλους τους ετούντες και στις αιτήσει που έχουμε λάβει πρέπει να σου πω πως οι περισσότερες, ε, από τις περισσότερες λείπουν κάποια στοιχεία πάντοτε, καμιά φορά ίσω σημασία και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να προσαρμοστεί κανείς σε ένα καινούριο σύστημα για την αναθεώρηση. Να σας πω ποιες είναι οι πρακτικές δυσκολίες. Υπάρχει μια σειρά ερωτήματα τα οποία προκύπτουν από το ίδιο το κόνσεπτ της μεμονωμένης άμεσης συμμετοχής σε κόμμα. Και ξεκινά από το εξή ερώτημα. Τι σημαίνει άμεσο μέλλον, να υπογράψει μια δήλωση. Πρέπει να υπάρχουν κάποια άλλα στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη. Επίσης, το πεδίο εφαρμογή για την εκπροσώπηση ε, στα περιφερειακά κοινοβούλια και κατά πόσο αυτό μπορεί να μπει ή όχι, γιατί δημιουργεί αυτό την ανάγκη να εξετάσουμε κάποια ζητήματα, για παράδειγμα αν υπάρχει και τοπικό ε, παράρτημα ε, εκτός από το περιφερειακό και πρέπει να σας πω πως εδώ είναι τεράστιος ο, ενδυνα... ο αριθμός ενδυνάμει μελών οπότε πρέπει να γίνει κάποια παλήθευση. Και είναι δύσκολο να εξασφαλίσει κανείς πως όλα τα κράτη-μέλη θα ακολουθούν την ίδια συνεκτική διαδικασία γιατί υπάρχει ε, και ο ορισμός σε επίπεδο κράτους μέλους για το τι αποτελεί περιφέρεια και τι είναι τοπικό επίπεδο. Δύσκολο και αυτό λοιπόν και έχουμε μετά και τα τρία στοιχεία που είπαμε, την περίπτωση που έχουμε συμμετοχή σε πολλά κόμματα, ε, μέλους ε, διαφόρων κομμάτων ή πολλαπλή ιδιότητα μέλους. Είναι δύσκολο αυτό να αποφασιστεί και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή προσπαθεί να μειώσει τη γραφειοκρατία, να μειώσει το διοικητικό βάρος για τους ετούντες, ακριβώ επειδή αλλάξαμε το σύστημα, έτσι ώστε οι ετούντες να μην υποχρεούνται να υποβάλουν μια φορά ε, προς την αρχή και μια φορά προς το Κοινοβούλιο τα ίδια έγγραφα. Εκεί έχουμε δουλειά να κάνουμε και αποτελεί και προτεραιότητα. Και στο μέλλον βέβαια θέλουμε να δούμε και πώς στην πράξη θα εφαρμόσουμε ε, το θέμα της χρηματοδότησης πολιτικών εκστρατιών εν ώψη και των εκλογών του 19 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε τρία σενάρια και είναι πάρα πολύ τεχνικό αυτό στο οποίο θα σταθώ. Έχουμε το πρώτο που θα το αποκαλέσω πολλαπλή ιδιότητα μέλους. Δηλαδή, έχουμε έναν ευρωβουλευτή που υπογράφει για δύο ευρωπαϊκά κόμματα. Και δεν ανήκει σε εθνικό κόμμα ευρωβουλευτή αυτός. Οπότε υπάρχει το εξή θέμα. Δηλαδή, το μετράμε δύο φορέ. Αν δεν το μετράμε δύο φορέ, σε ποιο τον μετράμε. Στο πρώτο που έχει δηλώσει. Στο πιο πρόσφατο. Και υπάρχει και η χρονική διάσταση που δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή, αν πούμε το πιο πρόσφατο πάντοτε, τότε Μπορεί ένας ευρωβουλευτής τη στιγμή της αίτησης προς την αρχή να θεωρεί πως εκπροσωπείται από ένα πάρτι και με, από ένα κόμμα και μετά αργότερα να βοηθήσει μέσω της παρουσίας του ή της ιδιότητας του μέλους κάποιο άλλο κόμμα να λάβει χρηματοδότηση. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά που προκύπτουν. Και βέβαια υπάρχει και η διασταυρούμενη ιδιότητα ε, μέλους. Τι σημαίνει αυτό. E λοιπόν, εδώ έχουμε την περίπτωση που έχουμε έναν ευρωβουλευτή ο οποίος αποτελεί μέλος ενός εθνικού κόμματος. Άρα έμεσα ανήκει στο Ευρωπαϊκό Κόμμα Α, αλλά υπογράφει δήλωση ότι ανήκει στο Ευρωπαϊκό Κόμμα Β. Οπότε είναι μια ουσιαστική διπλή ιδιότητα μέλους και αυτό δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στην ομοθεσία, Δηλαδή, ο Ευρωβουλευτής αυτός, γιατί η χρηματοδότηση μετράει στο Ευρωπαϊκό Κόμμα Α, άρα εκεί που είναι το εθνικό του κόμμα, αλλά όχι σε επίπεδο εκπροσώπησης. Οπότε και εδώ πάλι ε, είναι κάπως διτή η κατάσταση και δεν έχουμε ταύτιση εκπροσώπησης και χρηματοδότησης. Το οποίο σημαίνει ότι έχουμε μία τεχνητή διάκριση και δημιουργεί και το εξή ερώτημα, αυτό αντιστοιχεί στην επιλογή που έχει κάνει ο Ευρωβουλευτή ή όχι. Άρα λοιπόν είναι μια περίπλοκη ε, κατάσταση και προβλέπεται και τουλάχιστον σε επίπεδο χρηματοδότηση ξέρουμε πού θα τον μετρήσουμε. Και το τέλος είναι η πολυκομματική ιδιότητα μέλου. Κάτι το οποίο δεν ρυθμίζεται σήμερα στην Ομοθεσία. Έχουμε σε ένα εθνικό κόμμα δύο ευρωβουλευτές και οι δύο όταν έρχονται εδώ ανήκουν σε διαφορετικό ευρωπαϊκό κόμμα. Και αυτό επιτρέπεται με το τρέχον σύστημα. Δεν καλύπτεται από το 17 που είναι αυτό για τη διασταυρούμενη ιδιότητα μέλους. Άρα λοιπόν έχουμε μια ουσιαστική επικάλυψη πολιτικής τάση. Δηλαδή ανήκει στο ίδιο εθνικό κόμμα αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο εκπροσωπεί από δύο διαφορετικά κόμματα. Δηλαδή είναι ουσιαστικά ένας πολλαπλασιασμός, ένας επιπολασμός τάσεων μέσα στα κόμματα. Αυτό έχει συζητηθεί και δεν ε, βρίσκει κάποια λύση μέσα στο τρέχον σύστημα. Οπότε βλέπετε κι εσείς πως όλα αυτά τα θέματα συνδέονται με την ε, έννοια της ε, μεμονωμένης άμεσης συμμετοχής και πολιτικής συμμετοχής ή κομματικής ιδιότητας κάτι το οποίο καταργήθηκε και αν το καταργούσαμε μάλλον θα είχαμε λύσει το πρόβλημα, θα ήταν πιο εύκολο να διοικήσουμε το σύστημα και να το διαχειριστούμε. Κάποιοι το προτείνατε και σε τεχνικό επίπεδο ε, νομίζω έχετε δίκιο, σε περιφερειακό επίπεδο να σας πω ότι και αν το καταργούσαμε εκεί και πάλι εδώ θα ήταν πιο εύκολο να το διαχειριστούμε, πιο εύκολο να το υπελευθέρωσουμε και πιο εύκολο να το ελέγξουμε. Αυτά σε γενικές γραμμές για τα πρακτικά θέματα που προκύπτουν με την τρέχουσα νομοθεσία και σας ευχαριστώ πολύ που μας δώσατε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και μόλις έχουμε περισσότερα στοιχεία ή τεχνικές λεπτομέρειες που είναι χρήσιμες θα σας παρουσιάσουμε και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε πώς εφαρμόζεται ο κανονισμός και μάλιστα εν ώψη κάποιων μελλοντικών διαδικασιών αναθεώρησης που ενδεχομένως κάποια στιγμή θα προκύψουν. Ευχαριστώ. Πέντε συναδελφοί θέλουν να πάρουν το λόγο και εσείς μάλιστα. Okay, thank you. Uh, Ευχαριστώ. Μόρταν Μέσσερσμιτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Δύο θέματα. Πρώτον, για να καταλάβω μια ερώτηση προς τον κύριο Άνταμ για την ε, διπλή ιδιότητα μέλους. Ας πούμε το Σεπτέμβρη, το φθινόπωρο, υπογράφεις ε, ότι είσαι μέλος ενός πολιτικού κόμματος. Και αυτό ισχύει από την αρχή του επόμενου έτους. Αν είναι έτσι, αν θες να αλλάξεις πολιτικό κόμμα. Αν δεν είναι ανήκουστο, έχουμε συναδέλφους που πάνε από τη μία ομάδα στην άλλη. Πότε αρχίζει να ισχύει και τι επίπτωση έχει στη χρηματοδότηση. Αν θες για παράδειγμα να αλλάξει, να πας από το α στο β, θα πρέπει να υπογράψει για το νέο κόμμα, από ό,τι καταλαβαίνω, το Σεπτέμβριο. Αλλά ποιανού του σε μέλος τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Και πού πάει η χρηματοδότηση που σου αντιστοιχεί. Σε ρωτάω γιατί δεν κατάλαβα την παρουσίασή σα. Επίση, ένα θέμα που δεν έθεσαν οι δύο συνεισηγητές κατευθύνες γραμμές για την δαπάνηση των ενωσιακών πόρων. Αυτό είναι το θέμα, χωρίς να παραγνωρίζω τα άλλα τρία θέματα. Αυτά είναι τα θέματα που έχουν προκαλέσει συζητήσεις ε, στον τύπο και κριτικές. Πώς γίνονται αντιληπτοί αυτοί οι κανόνες που είναι κάπως γενικόλογοι Ποια είναι η προεκλογική περίοδος για ένα δημοψήφισμα για παράδειγμα. Με ποιο τρόπο τα μέλη ενό εθνικού κόμματο μπορούν να συμμετάσχουν στι δραστηριότητε ενό ευρωπαϊκού κόμματο. Να εξετάσουμε λοιπόν επίση αν αυτοί οι κανόνε θα μπορούσαν να είναι σαφέστεροι. Και για να έχουμε μια πλήρη θεώρηση και να αντιμετωπίσουμε τις κατηγορίες που αναφέρουν διάφορα μέσα ότι είναι αυθαίρετη η ερμηνεία αυτών των ε, κανόνων, να δημιουργήσουμε μια ομάδα εργασία που να εξετάσει το πώς έχουν εφαρμοστεί, πώς έχουν ερμηνευτεί οι κανόνες από όλα τα ευρωπαϊκά κόμματα τα τελευταία χρόνια για να δούμε ποιες είναι οι εγκεκριμένες πρακτικές. όταν έχουμε δυσκολίες με το πώς ορίζουμε τις προεκλογικές εκστρατείες, τα εθνικά κόμματα, αυτά που είπαν ήδη ομιλητέ. Τι είναι αποδεκτό για τη χρηματοδότηση. Τι έχει ισχύσει, τι έχει εφαρμοστεί την τελευταία πενταετία. Μία ομάδα εργασία με απόλυτη εμπιστευτικότητα, όπω έχουν κάνει και άλλε επιτροπέ, όπου τα μέλη να μπορέσουν να δούνε την ουσία για το πώ έχουν εφαρμοστεί αυτοί οι κανόνε σε όλα τα ευρωπαϊκά κόμματα και κατόπιν να κάνουν προτάσεις για σαφέστερους κανόνες στο μέλλον. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Οκτώ θέλουν το λόγο. Οπότε να μιλήσουν αρκετοί και να θυμάστε παρακαλώ τις ερωτήσεις τους. Helmut Scholz. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τις εισαγωγικές παρατηρήσεις των εκπροσώπων μας διαφόρων επιπέδων και ιδιαίτερα από το νέα φορέα. Είναι η πρώτη φορά που είχαμε δυνατότητα να ενημερωθούμε για τις απόψεις σας. Ένα από τα προβλήματα που συζητάμε σήμερα σχετίζεται με την καθυστέρηση που σημειώθηκε στην ε, δημιουργία του οργανισμού σας. Παρά το ότι η απόφαση λήφθηκε εδώ και αρκετά χρόνια. Το θέμα αυτό απέτυχε στην ουσία να το αντιμετωπίσει ο προηγούμενος εισηγητής του Κοινοβουλίου, την προηγούμενη θητεία. Για τα θέματα που συζητάμε σήμερα. Συζητάμε το δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών να συνέρχονται και να δημιουργούν πολιτικά κόμματα και σε ευρωπαϊκό θέμα. Αν συζητάμε λοιπόν εάν υπάρχουν ε, για παράδειγμα ε, δυνατότητες ε, μεμονωμένης συμμετοχή σε ευρωπαϊκό κόμμα ή και συλλογική συμμετοχή σε ενός εθνικού σε ένα ευρωπαϊκό κόμμα. Το θέμα είναι λοιπόν πώς θα εγγυηθούμε αυτό το δικαίωμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για όλους τους πολίτες. Δεύτερον, τα πολιτικά αυτά κακόματα, τα πολιτικά αυτά κόμματα, τα ευρωπαϊκά, μπορεί να αποτελούνται από εθνικά πολιτικά κόμματα που μπορεί να μην έχουν εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με βάση τον κανονισμό μας, τα ευρωπαϊκά κόμματα μπορούν να έχουν ε, μέλη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Μπορεί λοιπόν να μην είναι ευρωβουλευτές. να μην υπάρχουν ευρωβουλευτέ από τα κόμματα αυτά. Γι' αυτό βάλαμε στον κανονισμό ότι πρέπει να στηρίζονται και από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συμφωνώ ότι δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να υπογράφει ένα μέλος για πάνω από ένα Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα. Αυτό θα διευκρίνιζε την κατάσταση, αλλά παράλληλα δεν θα πρέπει να αυξηθεί το κατώτατο όριο. Γιατί για να τηρήσουμε τις δημοκρατικές αρχές θα πρέπει να αρκεί ότι υπογράφει ως μέλος αυτού του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος ένας Ευρωβουλευτής. Τρίτον, για να μην ε, μακρηγορήσω. Σε μια περίπτωση, διάφορα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε αυτή την τρέχουσα θητεία, επεχείρησαν να αμφισβητήσουν το δικαίωμα ύπαρξη και χρηματοδότηση κάποιων ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων για πολιτικού λόγου. Δυστυχώ, κάποια μέλη, τα μέλη αυτά μάλλον, δεν κατέδειξαν γιατί δεν ήταν σωστά τα στοιχεία που είχαν υποβάλει τα κόμματα αυτά. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Πήγα σε μια δίκη στην Ελλάδα της χρυσή αυγή. που με βάση την ελληνική νομοθεσία δεν έχει καταχωρηθεί ως πολιτικό κόμμα, αλλά εξακολουθεί να λαμβάνει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Άρα παρεμβαίνουμε σε εθνικές καταστάσεις. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, στην εθνική νομοθεσία, χρηματοδοτώντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και συγκεκριμένοι όταν συζητάμε τα συγκεκριμένα κριτήρια ποιες είναι οι προδιαγραφές για την δημιουργία και τη χρηματοδότηση ενός Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος. Τέταρτο. Το δικό μου κόμμα για παράδειγμα. Είναι μάλλον το μόνο κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα δεν είναι το, η ίδια συμμετοχή με την πολιτική ομάδα. Ενώ συμμετέχουν κόμματα που δεν συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να είναι δυνατό αυτό. Βεβαίω θέλουμε να αποκτήσουν ευρωπαϊκό χαρακτήρα τα πολιτικά κόμματα. Βεβαίω. Συμφωνώ με αυτό. Αλλά υπάρχει και το δημοκρατικό δικαίωμα των κομμάτων των χωρών της Ευρώπης να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ακόμη και αν δεν συμμετέχουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Και επιπλέον, πρέπει να συζητήσουμε ειλικρινά τα θέματα αυτά και να καλέσουμε τους εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων, Γενικούς Γραμματείς, Προέδρους, για να συζητήσουμε μαζί τους ποιοι θα πρέπει να είναι οι κανόνες για την μελλοντική συγκρότηση και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών θεμάτων. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με του συντονιστέ αύριο το πρωί. Θα το αποφασίσουμε λοιπόν. Για το άλλο θέμα που ανέφερε. νομίζω ότι ήδη αναφέρθηκε. Δεν υπήρξε καθυστέρηση. Ο κανονισμός που εγκρίθηκε το 2013 είχε και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για θέση σε ισχύ και δημιουργία των κομμάτων και ιδρυμάτων. Λοιπόν, η κυρία Καπαρντέλ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας και την διάθεσή σας να συζητήσετε τα θέματα αυτά για το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε με τη γνώμη μας ότι πρέπει να αναθεωρηθεί ο τρέχον κανονισμός το επόμενο φθινόπωρο. Νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή. Ε, απίφθηνα ήδη κατά την Ολομέλεια του Μαρτίου μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία πρότεινα μια σειρά αποτροποποίηση στον κανονισμό για να λύσουμε ορισμένα θέματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση. Είναι προφανές ότι πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός. Φυσικά το Κοινοβούλιο πάντα επιθυμεί όλες οι προτάσεις του να συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο δεν θα ήταν διατεθειμένο να τις υποστηρίξει όλες. Γι' αυτό νομίζουμε ότι η προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι. Ότι εφόσον δημοσιευτεί η πρόταση αναθεώρηση του κανονισμού θα πρέπει να επιδιώξουμε μια συνένεση μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων γιατί νομίζω ότι οι εκλογές του 2019 ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες εξελίξεις καθιστούν τις εκλογές αυτές πολύ σημαντικές για όλα τα κράτη-μέλη. Οι εκλογές αυτές θα είναι πολύ σημαντικές για το μέλλον της Ευρώπης. Γι' αυτό οι συνάδελφοι της Επιτροπής ΑΦΚΟ και εγώ έχουμε υποβάλει αρκετά επιχειρήματα για να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στην πρόταση της Κομισιόν και καταδείξαμε νομίζω γιατί πρέπει οπωσδήποτε φέτος να αναφερθεί ο κανονισμός. Ωστόσο θέλω να αναφέρω και ορισμένα στοιχεία των προτάσεων που ήδη αναφέρθηκαν αλλά θα ήθελα να τα υπενθυμίσω. Πρέπει να καταλάβουμε πολύ σωστά τα θέματα αυτά, το επίπεδο της συγχρηματοδότησης και των ιδίων πόρων. Γνωρίζουμε όλοι Οι συνδρομές των μελών ε, των κομμάτων δεν πληρώνονται επαρκώς και οι πόροι των πολιτικών κομμάτων μειώνονται συνέχεια. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να βοηθάει διάφορα πολιτικά κόμματα. Αλλά ορισμένοι μοιάζουν ότι να μην συμφωνούν. Εάν αλλάξουμε τους κανόνες, αυτό θα είχε επίπτωση σε μια σειρά από ε, λαϊκιστικές τάσεις που διαπιστώσαμε και εδώ και σε εθνικό επίπεδο. Η μήνυμου με προσώπηση. Αυτή η θεσμή είναι η πιο σημαντική της ευρωπαϊκής οικοδόμησης και δεν νομίζω ότι κόμματα που αποτελούνται από ένα, δύο ή τρία μέλη, όπου συμμετέχουν δηλαδή ένα, ένας, δύο ή τρεις ευρωβουλευτές, είναι σοβαρά. Πρώτον, ε, επίσης, συγγνώμη, η χρηματοδότηση των εθνικών ή τοπικών δημοψήφισμάτων είναι πολύ σημαντική, γιατί θέλουμε να προσεγγίσουμε όλο και περισσότερο τους πολίτες. Οπότε, επειδή ε, το δημοψήφισμα είναι πολύ χρήσιμο, πιστεύω ότι θα πρέπει να στηρίζουμε τέτοια δημοψηφίσματα. Επίσης, η μείωση της υποχρέωσης χρηματοδότησης για τα κόμματα περιλαμβάνεται ήδη στον υπάρχοντα κανονισμό. Ξέρουμε τι συνέβη πρόσφατα. Ήταν αποτέλεσμα διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο, ούτω ή άλλω αυτή η πρόβλεψη. Όμω επανερχόμεθα από αυτού, ακόμη και ξέροντα ότι δεν το θέλει το Συμβούλιο, γιατί ελπίζουμε ότι παρόλα αυτά θα το συζητήσουν τα κράτη-μέλη, θα το σκεφτούν. Γιατί σήμερα υπάρχει αύξηση των λαϊκιστικών τάσεων και των ακροδεξιών τάσεων. Πρέπει λοιπόν το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν την πρότασή μας. Και για να υπάρξει συμφωνία μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων για την αναθεώρηση λοιπόν του κανονισμού με τις προτάσεις αυτές που τις έχουν κάνει τα περισσότερα πολιτικά κόμματα νομίζω ότι κάθε ευρωβουλευτής πρέπει να έρθει σε επαφή με τις κυβερνήσεις και με τους εκπροσώπους μας ε, στο Συμβούλιο. Όλοι πρέπει να το κάνουν. Και να ολοκληρώσω με μία ερώτηση. Ελπίζω να μου απαντήσετε για να έχω άλλο ένα επιχείρημα για να υποβάλω στο Συμβούλιο στα πλαίσια των ενδεχομένων διαπραγματεύσεων. Ποια είναι λοιπόν αυτή η ερώτηση. Πώς πάει η αποτίμηση της ανάγκης αναθεώρησης. Είπαμε ότι θα έπρεπε να γίνει αναθεώρηση μετά από μια εκλογική θητεία. Αλλά επειδή έχει αλλάξει τόσο ριζικά η κατάσταση, επειδή έχει αυξηθεί τόσο πολύ ο λαϊκισμός, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουμε στάση. Αν θέλουμε το Κοινοβούλιο να μην χάσει την ε, αξιοπιστία του, πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν μια απάντηση στην ερώτησή μου και πιστεύω ότι θα πρέπει να εργαστούμε τάχιστα για την αναθεώρηση του κανονισμού. Ευχαριστώ πολύ. Τζο Λάινεν. Ήμουν ο πρώτος εισηγητής για αυτό το θέμα. 2003-2004. Και βλέπω με πολύ ενδιαφέρον τι συνέχεια είχε ο κανονισμός για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τι και να έχει τα οποία τότε δεν μπορέσαμε να τα δούμε και που τώρα θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θυμάμαι καλά το 2003-2004 τι συζήτηση κάναμε, τι είναι ένα Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα. Η Ένωση δεν είναι υποχρεωμένη να χρηματοδοτεί οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Αν κάποια ομάδα σε ένα κράτος μέλος έχει κάποια πολιτική δραστηριότητα και αν κάπου έχει μια διαμεθοριακή ε, διάσταση αυτή η δραστηριότητα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τη χρηματοδοτούμε. Στόχος μας ήταν να βοηθήσουμε πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να βοηθήσουν τους πολίτες της Ένωσης ε, να συμμετέχουν στις εκλογές και επίσης ε, και πολιτικές δυνάμεις που έχουν θέσεις έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο. Το 2003-2004 υπήρχαν τρία κράτη-μέλη όπου υπήρχαν πολύ μικρά κόμματα στην κυβερνητική πλειοψηφία. Και γι' αυτό λέει ακόμη ο κανονισμός ότι αρκεί ένας ευρωβουλευτή. Αυτή ήταν η αιτία. Μας ε, εξεβίασαν τρει κυβερνήσεις που αλλιώ δεν θα είχαν συμφωνήσει. Και χρειάστηκε να πούμε εντάξει φτάνει ένα ευρωβουλευτή. Και όντω συμφωνώ ότι είναι πολύ λίγοι. Λίγος ένας. Δεν να χρειάζεται δούμε οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Χρηματοδοτούμε πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να συμμετάσχουν σε ευρωεκλογέ και οι οποίες επιτυχάνουν να εκλέξουν ευρωβουλευτές. Πρέπει λοιπόν να ανέβει το κατόφλιο, όχι μόνο ένας. Αυτό είναι ο στόχο όταν χρηματοδοτούμε ε, πολιτικές δραστηριότητες, γιατί δεν είμαστε μόνοι που χρηματοδοτούμε. Υπάρχουν ε, υπάρχουν διάφορα ιδρύματα που χρηματοδοτούν πολιτική δραστηριότητα. Δεν είναι στόχο μα να χρηματοδοτούμε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Ο κύριο Άνταμ τα παρουσίασε πολύ σωστά. Τι καταχρήσει έχουμε διαπιστώσει. Διπλή ιδιότητα μέλου, ε, ε, πολλαπλή ιδιότητα μέλους και ε, διασταυρούμενη ιδιότητα μέλου. Πολύ δημιουργικά όλα αυτά, αλλά είναι σαφέ ότι είναι καταχρήσει και πρέπει να σταματήσουν. Δεν είναι δυνατόν να μετράει δυο φορέ κάποιο. Ω βουλευτή και ω κόμμα, μία φορά μετράει ο καθένα. Μία φορά μετράει ο καθένα. Πρέπει λοιπόν να κλείσουν αυτέ οι τρύπε, αυτά τα κενά. Σημειώθηκε όμω πρόοδο. Στον πρώτο κανονισμό δεν ήταν δυνατόν να χρηματοδοτηθεί η προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογέ. Επίσης και για ευρωπαϊκά δημοψηφίσματα υπάρχει δυνατότητα και αυτά εκλογέ είναι και αναφερθήκατε και στη διαδικασία του επικεφαλή των ψηφοδελτίων και αυτό είναι καινούργιο. Αυτό είναι τμήμα των πολιτικών εκστρατιών και της ε, συζήτησης με την κοινή γνώμη ενώψη ευρωεκλογών. Η χρηματοδότηση λοιπόν των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων πρέπει να γίνει με αυτούς τους στόχους. Έχουμε λοιπόν τώρα ε, μια ευρεία γκάμα πολιτικών κομμάτων που χρηματοδοτούνται. Αυτό είναι καλό. Από την αρχή είχαμε τονίσει ότι δεν είναι πρόβλημα αν κάποιο είναι επικριτικός έναντι της Ευρώπη. Και μετά στο Κοινοβούλιο είδαμε άτομα όχι απλώς επικρίνουν, αλλά θέλουν να καταστρέψουν την Ένωση. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση, εάν και κατά πόσο θα πρέπει να χρηματοδοτούμε δυνάμεις που δεν θέλουν να τροποποιήσουν την Ένωση, αλλά που απορρίπτουν σαφέστατα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί θα πρέπει η Ένωση να χρηματοδοτεί πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να την καταστρέψουν. Είναι μια κόκκινη γραμμή που δεν την τραβήξαμε τότε. Ίσως ήταν πρόωρο να την έχουμε τραβήξει την κόκκινη γραμμή από τότε αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει και αυτό. Ορισμένοι δεν απορρίπτουν απλώ την Ένωση, αλλά και τι αξίε τη Ένωση. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, υπήρξε μια απόφαση του, του... του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου που είναι πολύ γενναιόδορη όσον αφορά το κατά πόσο επιτρέπεται να λειτουργεί ένα κόμμα. Είπε ότι ακόμη και το ναζιστικό κόμμα δεν το απαγορεύουμε. Αλλά εάν ε, αντιμετωπίζει με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο τις αξίες μας, πρέπει και να το χρηματοδοτούμε. Πρέπει να υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο να επιτρέπεται να λειτουργεί ένα κόμμα και στο να λαμβάνει δημόσια χρηματοδότηση. Αναφέρθηκαν παραδείγματα, όπου θα πρέπει ακριβώς να εξετάσουμε. Μα πού δίνουμε τα λεφτά μας. Αν είναι κάποιοι κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών, αυτός είναι ο πλουραλισμός που θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε. Επιτρέπεται στη δημοκρατία. Αλλά πρέπει να το χρηματοδοτούμε και από πάνω. Ευχαριστώ κυρία Νταϊάν Τζέιμς, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω κάποιες παρατηρήσεις. Θα, αναφερθώ ακριβώ σε αυτές. Ελπίζω όλοι στην αίθουσα να δέχονται ότι το πολιτικό περιβάλλον μεταβάλλεται. Κανείς δεν είχε προβλέψει ότι η Γαλλία θα έχει ηγηθεί σε αυτό το τομέα και το πώς αναδύθηκε ο Μακρόν και το κόμμα του. Είναι ενδιαφέρουσα πτυχή, έτσι δεν είναι. Πώς εντάσσεται αυτό στις επόμενες ευρωεκλογέ. Υπάρχει ένα κόμμα που φεύγει από μια χώρα που φαίνεται να αποτελείται διακομματικά και πώς θα συμμετάσχει στην κατανομή των εδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά εμφανίζονται και κινήματα, πολιτικά κινήματα αυτό αναγνωρίζεται περισσότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο από τι άλλε χώρε. Αλλά υπάρχουν κάποιε ενδείξεις και κάποια μαθήματα που μάθαμε από αυτό. Το πιο σημαντικό είναι η φύση της μη αποκάλυψης της άμεσης ε, συμμετοχής σε ένα πολιτικό κόμμα και της κατευθύνσεως. Αυτό θα πρέπει να αποκαλύπτεται. Αν είναι πίσω πόρτα ούτω ώστε να δίνουμε μεγαλύτερη πυγμή σε ένα πολιτικό κόμμα τότε αυτό αντιβαίνει το δημοκρατικό ήθος και το θέμα της διαφάνειας. Το τρίτο σχόλιο, το θέμα της συλλογή χρηματοδότησης, ε, crowdfunding, νέα μέθοδος χρηματοδοτήσεως πολιτικών κομμάτων. Και είχαμε μια περίσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, 80.000 δωρητές σε 24 ώρες έδωσαν ένα σημαντικό ποσό χρημάτων σε μια πολιτική εκστρατεία. Τώρα, το να προσπαθήσει κανείς να εντοπίσει τους 80.000 αυτού ανθρώπους ε, ήταν κάτι ανέφικτο. Αλλά η νομιμότητα των χρημάτων που δωρήθηκαν πρέπει να εξεταστεί και αν θέλετε χρειάζεται ένα επίπεδο αστυνόμευσης, ούτως ώστε ε, αυτή η προσέγγιση να μην επηρεάζει αρνητικά τις εκλογές και την ε, εκπροσώπηση. Τέταρτο σημείο. Τίνω να συμφωνήσω με κάποια σχόλια για την απαγόρευση κάποιων κομμάτων. Είναι ενδιαφέρον αυτό που ακούσαμε. Ακούσαμε μόνο την απαγόρευση κομμάτια ακροδεξιά. Θα ήθελα να ενθαρρύνω και κάτι άλλο. Άκουσα ότι οι Γερμανοί σκέφτονται την απαγόρευση και τη άκρα αριστερά, διότι είναι αρκετά επικίνδυνη και από την εκείνη την πλευρά, όσο είναι και από τη δεξιά πλευρά. Ε, είναι ένα ε, τομέα όπου εκεί δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που με επιτρέψατε να παρουσιάσω τα σημεία μου και προσπάθησα να είμαι συνοπτική. Ε, ο κύριος Τέρη Καμπέρας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να κάνω μία πολύ γενική ερώτηση. Είμαστε κατά των ευρωπαϊκών κομμάτων. Είμαστε υπέρ. Όλοι θα απαντήσουν ότι είναι υπέρ. Αλλά ανάλογα με το πώς το αντιμετωπίζει κανείς, καταλαβαίνουμε αν είναι κανείς πραγματικά υπέρ ή όχι. Αν θέλει να τα απαγορεύσει σε τελευταία ανάλυση ή να καταστήσει αδύνατη τη λειτουργία τους. Είναι θέμα δημοκρατίας. Καταλαβαίνω καλά το ότι τα μεγάλα κόμματα θέλουν να γίνουν μεγαλύτερα. Αυτό το καταλαβαίνω πολύ καλά. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί τα μεγάλα κόμματα Θέλουν να απαγορεύσουν και να εξαφανίσουν τα μικρότερα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Γιατί. Εγώ είμαι υπέρ των ευρωπαϊκών κομμάτων και εκφράζομαι ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, EFA, και είμαι και υπέρ λοιπόν των μικρών κομμάτων. Αλλά πρώτα απ' όλα είμαι υπέρ των, και πάνω απ' όλα, είμαι υπέρ των ευρωπαϊκών κομμάτων. Θέλουμε, μάλλον, διαπιστώνουμε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι οι συμπολίτες μας από την Ευρώπη, ότι απομακρύνονται. Και μετά παίρνουν αποφάσεις κατά των πολιτών που ανήκουν στα μικρά κόμματα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Είμαι απολύτως κατά βεβαίως. Αλλά είμαι υπέρ ότι πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι ε, επί της λειτουργίας των πολύ αυστηρή έλεγχη. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει διασταυρούμενη ιδιότητα μέλου, δεν είναι δυνατόν ένα βουλευτή να συμμετέχει σε δύο κόμματα. Αυτά είναι ευλακίε. Υπάρχουν καταχρήσεις, φυσικά υπάρχουν. Θέλουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν κόμματα τα οποία ε, έχουν κάνει και οικονομικές ατασταλίες. Αυτά πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αλλά κάτι ακόμη για τον αριθμό ευρωβουλευτών. Ένα ευρωπαϊκό κόμμα είναι ένα δίκτυο πολιτικών και πολιτών που έχουν μέλη σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο ή και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό στηρίζουμε ή δεν στηρίζουμε. Το ότι χρειάζεται μόνο ένας ευρωβουλευτής, αυτό δεν είναι το σημαντικό. Ένας ή εκατό, το δίκτυο υπάρχει ή και δεν υπάρχει. Αυτό πρέπει να ελέγξουμε, αν υπάρχει ή όχι, αλλά όχι τους βουλευτές. Και για μένα είναι αδιανόητο. Ενώ υπάρχει ευρωβουλευτής να μην λάβει καμία χρηματοδότηση. Αυτό είναι απίστευτο. Γιατί να υφίσταται διακρίσει. Ακόμη και αν είναι μικρή η ομάδα του. Και εάν λάβει την αναγκαία χρηματοδότηση, μετά μπορεί να μπουν και άλλοι ευρωβουλευτέ. Και αν γίνουν 2-3% τότε θα πάρουν περισσότερη χρηματοδότηση. Το καταλαβαίνω, μαθηματικά είναι αυτά. Αλλά δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τους πολίτες που ανήκουν στα μικρότερα κόμματα. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τους συναδέλφους που έχουν εκλεγεί από τους συμπολίτες μας. Οι οποίοι είναι καλοί, εξίσου καλοί και δημοκράτες όπως και εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Χέραλτ Άνεμαντς και ο κ. Ο πρώτος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ομάδα μου, όπως είπα και την άνοιξη στο Στρασβουργό, η ομάδα μου εξετάζει όλα τα μέτρα εκείνα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να εκαθαριστεί το σύστημα έγιναν κάποιες χρήσιμες προτάσεις. Μιλώ σαν Ευρωβουλευτής που επί 30 χρόνια ήταν Ευρωβουλευτής και ανήκει πάντα στο ίδιο Εθνικό Κόμμα και πάντα ήταν σαφής η εκλογή μου, ξεκάθαρη και δεν κατανοώ γιατί έχουν περιπλακεί τα πράγματα. Αποφασίζει ένα Εθνικό Κόμμα ε, ποιον θα έχει μέλος. Δεν μπορεί να έχεις άλλα μέλη του κόμματος να γίνονται μέλη άλλων κομμάτων τα κόμματα πρέπει να το προσέξουν αυτό. Ήμουν υπέρ γενική διορθώσεω τη καταστάσεω και καθάριση και θα παίξω το ρόλο που μου αρμόζει. Αναφέρθηκε και το να ε, εξετάσουμε και τις περιπτώσεις αυτές που τα κόμματα να έχουν πάνω από ένα μέλος. 25 μέλη, όχι. Αυτός ο αριθμός ε, είναι πολύ ψηλός. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κανείς ε, ανθρώπους να σχηματίσει μια ομάδα. Τρία μέλη, επτά μέλη, αυτό μπορεί να συζητηθεί, μπορείς να υπογράψεις μια φορά, αν δεν ανήκεις σε εθνικό κόμμα, μια φορά μπορείς να υπογράψεις, είναι ένα απλούστατο σύστημα. 30 χρόνια ήμουν ευρωβουλευτής, όπως σας είπα, στο σύστημα το βελγικό χρηματοδοτήσεως πολιτικών κομμάτων, ε, ποτέ με την ιδιότητά μου σαν ευρωβουλευτής δεν είδα πρόβλημα. Θα ήθελα να δω να, έχει, να υπάρχουν δύο κράτη στο Βέλγιο. Είμαι κατά του βελγικού κράτους. Παρ' όλα αυτά έχει χρηματοδοτηθεί επί 30 χρόνια το κόμμα μου από το βελγικό κράτος επί 30 χρόνια. Δεν είναι επειδή είμαι κατά του κράτους αυτού ότι δεν χρηματοδοτήθηκα. Δεν είμαι υπέρ ή κατά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένος κάποιος να ανεμίζει ευρωπαϊκή σημαία και να είναι υπέρ τη φεντεραλιστική Ευρώπη να χρηματοδοτηθεί. Εάν εκλέγεται κάποιο, εκπροσωπεί λαό, κόσμο. Νομίζω ότι πάμε πολύ μακριά αν οι βασικοί επηρεαστούν οι βασικές ιδέες, αν επηρεάζονται οι βασικές ιδέες ενός κόμματος από επιδοτήσεις, από χρηματοδότηση. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ όσον αφορά την εκαθάριση του συστήματος, τότε είμαι έτοιμος και εγώ να συμβάλλω με την προσπάθειά μου. Ο επόμενος παρακαλώ. Ο κύριος Σελίμωβιτς, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και όλους τους προλαλήσαντες, όπως επίσης και όλους τους συναδέλφους οι οποίοι συζήτησαν τα θέματα αυτά και κάποιος κάνει το, ε, την εξή ερώτηση. Το αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Τα αγαπάμε αυτά τα κόμματα. Ναι, ναι, και θα υπάρχουν και στο μέλλον και θα έχουν και περισσότερη δράση ε, στο μέλλον και πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό αυξάνουμε την νομιμότητα, την νομιμοποίηση μάλλον των ε, ε, ευρωπαϊκών οργάνων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτά τώρα συζητάμε. Είδαμε πώς προχωράει η διαδικασία του επικεφαλής ψηφοδελτίου, όπου η Ευρωπαϊκή πολίτες μπορούν όχι μόνο να εκλέξουν ποιοι θα τους, ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και ποιο θα ηγηθεί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι καταλήγουμε σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την νομιμοποίηση της δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τα κόμματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως ένας τρόπος ακριβώς να αυξήσουμε αυτή την νομιμοποίηση στα μάτια του πολίτη. Πιστεύω λοιπόν πως είναι πραγματικά απαραίτητη η αναθεώρηση έχει φτάσει την κατάλληλη στιγμή και θα ήθελα να στηρίξω τρία από τα σημεία που έχουμε ε, στην επιστολή που έστειλαν και υπέγραψαν ε, οι επικεφαλής τριών ε, πολιτικών κομμάτων, συμπεριλαμβάνουμε και τους φιλελεύθερους που δεν είναι εδώ, η μείωση κατά 15% ναι, αύξηση της ε, εκπροσώπησης ώστε να είναι τρεις τουλάχιστον ευρωβουλευτές, γιατί βέβαια τα ατομικά κόμματα νομίζω είναι κάποιο περίεργο μόρφωμα και θα πρέπει βεβαίως να σταθούμε και στην πρόληψη της πολλαπλής κομματικής ε, ιδιότητας για τους ευρωβουλευτές. Ένα τέτοιο κανονισμό θα πρέπει να διευκρινίζει και ένα πολύ δύσκολο ερώτημα που έθεσαν κάποιοι ε, συνάδελφοι. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η περίφημη κόκκινη γραμμή. Εγώ πιστεύω πως τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα θα πρέπει πάντα να συμμορφώνονται και να σέβονται τις αρχές που έχουμε στο άρθρο 2 της Συνθήκης, στην Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και επίσης πως οποιοδήποτε κόμμα ε, ε, κάνει ε, δηλώσεις ρατσιστικές, μυσαλόδοξες κτλ. δεν θα πρέπει να χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Και αυτό βεβαίως σημαίνει και μία κόκκινη γραμμή εδώ και ξέρω Πώ δεν είναι εύκολο να βρει κανεί ποιε είναι αυτέ οι κόκκινε γραμμές και με ποιου κανόνε θα χαραχθούν, αλλά πρέπει να γίνει, είναι σημαντικό. Και αυτή η αναθεώρηση θα πρέπει να το σκεφτεί. Γιατί, Γιατί είδαμε πως τα κόμματα αυτά έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται στην Ευρώπη ε, ένα ε, ξέσπασμα, μια έκρηξη υποστήριξη προς τα κόμματα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ας τραβήξουμε λοιπόν μια γραμμή και ας αποφύγουμε την πολύ δύσκολη ε, κατάσταση όπου χρειάζεται κάποιος ε, να απομακρυνθεί εφόσον έχει καταλάβει την εξουσία που όντως εκεί υπάρχει πρόβλημα. Οπότε εκεί διευκρινήσεις παρακαλώ, καταλαβαίνω πως είναι δύσκολο αλλά νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Θα ήθελα επίσης να ακούσω και κάποια παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες από τους προσκεκλημένους μας για το θέμα αυτό. Και ε, επειδή αυτή τη στιγμή τρέχει και μια άλλη συνεδρίαση, σα ζητώ συγγνώμη, πρέπει να αποχωρήσω, αλλά θα ήθελα να εξασφαλίσω και ε, να, να σας ε, πω, αγαπητοί προσκεκλημένοι, πως εμένα θα μου σημειώσουν τις απαντήσεις και θα τις λάβω δεόντως υπόψη. Ωραία. Μείνανε λοιπόν και 20 λεπτά για τους προσκεκλημένους για να απαντήσουν. Δεν ξέρω με ποια σειρά θέλετε να μιλήσετε. Ράινερ, εσύ πρώτος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για την ευγενική παράκληση. Να αντιληφθούμε ότι δεν είναι πολύ καλό το κείμενό μας μέχρι τώρα. Αλλά μόνο και μόνο το γεγονός ότι πρέπει να αποτιμηθεί το 18. Εάν αρχίσουμε το Γενάρη, θα τελειώσουμε το Δεκέμβρη, δηλαδή πέντε μήνες πριν από τις εκλογές. Οπότε όλο αυτό το θέμα θα είναι θέμα της προεκλογικής εκστρατείας. Αυτό είναι παλαβό. Δεύτερον, το θέμα δεν είναι ο καλός ο κακός ο άσχημος. Δεν είναι ποιος είναι καλός ως κόμμα δηλαδή και ποιος είναι κακός. Ναι, ναι, και εγώ διάβασα τι είπαν στην Καρζούη δεν είναι τόσο απλές προϋποθέσεις όπως αναφέρει το δικαστήριο. Έχει να κάνει και με το τι επιτυχία έχει το κόμμα. Πρέπει να διαβάσουμε σωστά την απάντηση. Και επιπλέον δεν είναι το θέμα ότι θέλουμε να ευνοήσουμε τους ε, μεγάλους και όχι τους μικρούς. Οι μικροί σε όλα που κάνουμε ευνοούνται. Για τον λόγο χρόνο ομιλίας για παράδειγμα υπάρχει ένα ε, κατώτατο όριο για όλους. Όλοι όλοι οι μικροί ευνοούνται και στις διαπραγματεύσεις συμμετέχουν δύο από του μεγάλους και ένας από τους κάθε μικρό. Πρέπει λοιπόν να προσέχει τι λέει ο συνάδελφο Τέρι Κάμπρα. Το θέμα είναι πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν οργανώνουμε δηλαδή πλέον, δεν θέλουμε να οργανώσουμε πλέον αυτή την κατάχρηση δημοσίων πόρων. Θέλουμε να αποφύγουμε την κατάχρηση. Γι' αυτό θέλω να πούμε. Όποιος αλλάζει κόμμα. Θα μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω. Αλλά όχι πολύ παραπάνω. Δηλαδή, ας, εάν ως μεμονωμένος βουλευτής φεύγω από ένα κόμμα, δεν μπορώ να φτιάξω καινούριο. Αν δεν έχω και μερικούς άλλους. Ένα, δύο ή τρεις. Δηλαδή μπορώ να συμβάλλω μόνο μια φορά στη δημιουργία κόμματο. Μετά μπορώ να πάω σε άλλο κόμμα, στο οποίο να υπάρχει ήδη. Αν πάω σε αυτό το άλλο θα πάρουν αυτοί λίγο περισσότερα χρήματα, αλλά δεν μπορώ εγώ με κάποιους άλλους, για παράδειγμα, που και αυτοί έχουν φύγει από τα κόμματα στα οποία είχαν συμμετάσχει, να ιδρύσουμε κι άλλο. Αυτό είναι το βασικό. Η συμπληρωματοδότηση είναι προφανής. και ότι θα πρέπει να είναι πάνω από ένας ευρωβουλευτής και γι' αυτό και αυτό είναι σαφές για μένα. Αλλά πρέπει να προσέξουμε. Να μην κάνουμε το ίδιο λάθος που κάναμε και το εκλογικό δικαίωμα όπου παραφορτώσαμε το θέμα και γι' αυτό έχει κολλήσει. Σήμερα επίσης κάναμε το λάθος. Επειδή δεν λύσαμε το θέμα των εδρών, τώρα συζητάμε για διεθνικά ψηφοδέλτια. Δεν έχει λοιπόν έννοια να πούμε πάρα πολλά επιθυμητά και ενδεχομένω θετικά. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι τώρα αμέσως μετά τις επόμενες εκλογές θα πρέπει να κάνουμε μία εκβάθρον συζήτηση για να δημιουργήσουμε ένα νέο σύστημα πριν τι εκλογές του 2024. Νομίζω ότι η βασική έλλειψη είναι η εξή. Συνδέουμε το παρόν με το μέλλον με αυτά τα οποία πληρώνουμε τώρα. Αν αντίθετα θα έπρεπε να κοιτάμε προ τα πίσω. Πόση επιτυχία έχει στις εκλογές. Και πρέπει να το συνδέουμε τον αριθμό των ψηφοφόρων. Όχι με τον αριθμό των ε, εκλεγμένων οι πολιτικές ε, ομάδες λαμβάνουν χρηματοδότηση με βάση τον αριθμό των μελών τους. Τα κόμματα θα πρέπει να λάβουν χρηματοδότηση με βάση τον αριθμό των ψηφοφόρων τους. Και μετά ο κάθε ευρωβουλευτής μπορεί να πάει όπου θέλει. Να, εγώ είμαι Γερμανός, μπορώ να πάω και σε ένα εστονικό κόμμα, αν θέλω μετά. Αλλά η φόρμουλα που πρέπει να επιλέξουμε θα είναι sui generis γιατί το δίκαιο των κομμάτων είναι διαφορετικό. Στη χώρα μου, για παράδειγμα, ορισμένα, τα κόμματα κάνουν ορισμένες, έχουν κάποια καθήκοντα, τα οποία δεν μπορούν να κάνουν ενώσεις και αντίστροφα. Πρέπει να υπολογίζουν, για παράδειγμα, για τα κόμματα, οι αρχές, τι δραστηριότητες έχει, και τι χρηματοδότηση παίρνει από ιδιώτε ή από τι συνδρομέ των μελών. Και αυτά τα κόμματα που έχουν επαρκή χρηματοδότηση από αυτά δεν παίρνουν ε, χρηματοδότηση δημόσια. Έχουμε 500 εκατομμύρια πολίτε. Θα έχουμε γύρω στα 300 εκατομμύρια ψηφοφόρου. Από αυτού ε, ψηφίζουν ε, γύρω στο 50%. Έχουμε λοιπόν 150 εκατομμύρια. Και έχουμε 32 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή δίνω περίπου 30 λεπτά ανά ψηφοφόρο. Μπορείτε λοιπόν να υπολογίζετε με αυτόν τον τρόπο τι πρέπει να πάρει κάθε κόμμα. Εάν το κόμμα του κυρίου Τερικάμπρας πει ότι θέλω να φτιάξω ένα αδελφό κόμμα στην ε, Πορτογαλία, τότε πρέπει να πει το κόμμα του κυρίου Τερικάμπρας θα πανίσω χρήματα γι' αυτό. Εάν ένα κόμμα διαλύεται στην Αγγλία πρέπει να τα βοηθήσουμε. Μία χώρα, για παράδειγμα, είναι σε διαδικασία ένταξης. Θέλω να φτιάξω ένα αδελφό κόμμα εκεί. Θα πρέπει να μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Εάν οι κανόνες μας είναι καλύτεροι, τότε δεν χρειάζεται να ελέγχουμε τόσο αυστηρά. Απλώς θα πρέπει να θέσουμε μία-δύο κόκκινες γραμμές. Θα πρέπει να περιοριστούμε σε αυτά τα οποία είναι διατεθειμένοι τώρα να κάνει η Κομισιόν και μετά να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία. Αμέσως μετά τις επόμενες ευρωεκλογέ που θα είναι η κατάσταση πιο χαλαρή. Εντάξει, το θέμα αυτό ε, έχει απασχολήσει το Συμβούλιο επί 15 χρόνια, όπως είπε και ο συνάδελφος ε, Λάινεν. Να δούμε πολύ προσεκτικότερα ποια είναι η κουλτούρα για τα κόμματα σε κάθε κόμμα και να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική κουλτούρα, ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Η Ουλρίκε. Ναι, και εγώ συμφωνώ με ορισμένες από τις ιδέες του συναδέλφου Βίλαντ. Νομίζω ότι η Κομισιόν πρέπει να επικεντρωθεί στο να κλείσει τα κενά και στα σημαντικότερα θέματα. Αυτό έχει έννοια. Και αυτό μπορεί να γίνει σχετικά σύντομα. Τα υπόλοιπα θέλουν περισσότερο χρόνο. Και αυτή είναι η δική μου πρόθεση. Και αναφέρουμε και ένα άλλο σημείο. Για τους ίδιους πόρους. Αυτή η μείωση, η πρόταση που υπάρχει εδώ από το Κοινοβούλιο, πρέπει να συμπεριληφθεί. Και αυτή τη θεωρώ πολύ σημαντική. Εγώ θεωρώ σαν Φεβίλαντ ότι μπορούμε ως κοινοβούλιο να εκφράσουμε τις επιθυμίες μας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να εκφράσουμε τις επιθυμίες μας. Η ιδέα που αναφέρθηκε, η ιδέα που είπατε, ότι η χρηματοδότηση των κομμάτων θα πρέπει να μελετά τι στήριξη έχουν τα κόμματα στο παρελθόν. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε, αν έχει έννοια. Αλλά καταλαβαίνω τι εννοείται. Ένα κόμμα, όπως διαπιστώσαμε τα τελευταία χρόνια, ένα κόμμα λέει βεβαίως να πάρουμε αυτή τη χρηματοδότηση και θα ξεκινήσουμε να λειτουργούμε και κανείς δεν ξέρει προς ποια κατεύθυνση θα πάει. Αυτό που είπατε εσείς ότι τα κόμματα πρέπει να έχουν μια ε, φιλοευρωπαϊκή στάση. Πρέπει να ε, βασίζονται στις βασικές αρχές της χάρτας. Και έτσι μπορούμε να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ εκείνων που όπως λέει ο κύριος ε, ε, Άνεμανς που έφυγε θα πρέπει να καταλάβουν κόμματα όπως το Φλαμπ Μπελάν και το ENF δεν μπορούν να ζητούν χρηματοδότηση όταν στρέφονται κατά των αρχών εκείνων που τους ε, χρηματοδοτούν. Βεβαίως, η αναφορά στα θεμελιώδη δικαιώματα για τη χάρτα είναι σημαντική. Τώρα για τον αριθμό των βουλευτών, των ευρωβουλευτών και ποιοι άλλοι θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την ίδρυση ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Ο συνάδελφο Τέρι είναι μέλο τη ομάδα μου. Καταλαβαίνω ότι η Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία ως λειτουργία έχει να κάνει με τη διαφορετική διάσταση των κρατών μελών. Στη χώρα μου η χώρα μου είναι το 1 δέκατο της Γερμανίας. Υπάρχουν πολλές χώρες όπου υπάρχουν και μειονότητες, γλωσσικές μειονότητες, όπου οι περιφέρειες ορίζονται διαφορετικά. Να πούμε τώρα λοιπόν ότι δεν θέλουμε να μην αρνηθούμε την νομιμοποίηση ενός τοπικού εκλεγμένου. Ξέρετε, μεταξύ του Λουξεμβούργου και της Γερμανίας και της Πολωνίας η διαφορά μεταξύ ε, τοπικών εκλεγμένων και περιφερειακών εκλεγμένων είναι πολύ ε, μεγάλη. Δεν μπορούμε να τα κρίνουμε όλα με τα ίδια κριτήρια. Και αν ε, συμπεριλάβουμε και τα κριτήριο της φιλοευρωπαϊκής τάσης, τότε μπορούμε να περιοριστούμε σε ένα ή δύο μόνο ευρωβουλευτές. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Ουλρίκη. Διτιέ, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να μπορώ να συμμετάσχω στην πολιτική συζήτηση που είναι αυτή που πρέπει να κάνετε εσείς, αλλά νομίζω ότι εμείς ως γραμματεία θα ασχοληθούμε με τις προτεραιότητες τις οποίες εξέφρασαν οι περισσότεροι εδώ. Δηλαδή, συγχρηματοδότηση, μείωση αυτής, αντιπροσωπευτικότητα ελάχιστη με έναν ευρωβουλευτή ή περισσότερους, το θέμα της διασταυρούμενης ε, κομματικής ιδιότητας, να ξεκινήσω με μια μικρή παρατήρηση για τις διάφορες συζητήσεις. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι που θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη, που είναι οι εθνικοί κανόνες, μια και μιλάμε για χρηματοδότηση εθνικών κομμάτων ή προεκλογικών εκστρατιών ή δημοψηφισμάτων, γιατί πολλές φορές σε, ευρωπαϊκή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε το επιτρέπουμε είτε όχι, τα πολιτικά κόμματα μπορούν να συμμετέχουν σε ε, δημοψηφίσματα. Ε, παρόλο που στη νέα νομοθεσία δεν έχουν αυτό το δικαίωμα ούτε με δική τους χρηματοδότηση. Οπότε αυτά θα πρέπει να τα δούμε σε συνδυασμό με τους εθνικούς κανόνες και να δούμε τα όσα διαπιστώσαμε εκεί, για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους ε, η σχετική αρχή στο Ηνωμένο Βασίλειο παρακολουθεί πολύ στενά πώς εξελίσσονται όλα τα θέματα αυτά. Δεν μπορούμε λοιπόν τα θέματα αυτά να αντιμετωπίσουμε με εύκολες λύσεις, αλλά θα πρέπει να βρούμε αυτές που θα μας επιτρέψουν να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε μελλοντικά προβλήματα εμφανιστούν. Επίσης, υπάρχει η αρχή της αυτορύθμισης, του αυτοπεριορισμού. Μιλώ, για παράδειγμα, για το δικαίωμα του συνέρχεστε και συνεταιρίζεστε και αυτό είναι ένα δικαίωμα των πολιτών που μπορούν να δημιουργήσουν ένα πολιτικό κόμμα και με τον τρόπο αυτό μπορεί να εκφράσουν ε, την πολιτική βούληση των Ευρωπαίων πολιτών. Δηλαδή τρία-επτά άτομα δύσκολα μπορούν μαζί να συνδυαστούν έτσι ώστε να καλύψουν αυτό το στόχο και να αναγνωριστούν ως πολιτικό κόμμα στην Ευρώπη και να χρηματοδοτηθούν. Οπότε ε, θα πρέπει να βρεθεί κάποιο σημείο ισορροπίας. Μιλάμε για μια αυτορύθμιση ουσιαστικά που είναι και το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ κυρία Γιώχανσον. Θα ήθελα κι εγώ να σας ευχαριστήσω για την πολύ χρήσιμη συζήτηση. Γιατί αυτή τη στιγμή κοιτάμε τις τροπολογίες για την νομοθεσία και θα μας βοηθήσετε στο να διατυπώσουμε όλα τα θέματα αυτά σε ένα νομικό κείμενο και αποδεικνύει πόσο περίπλοκο είναι το θέμα, πόσες πολλές είναι οι διαστάσεις που πρέπει να δούμε και να αντιμετωπίσουμε. Καταρχήν, το χρονοδιάγραμμα είναι πάρα πολύ φιλόδοξο. Είπαμε οι δύο συνομοθέτες να συμφωνήσουν μέχρι την άνοιξη του Άρα λοιπόν θα πρέπει αμέσως να κάνουμε τις αλλαγές που είναι απαραίτητες και να γίνει και μια ευρύτερη συζήτηση αργότερα. Θέλω λοιπόν να στηρίξω τις προτάσεις σας έτσι ώστε τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και να ε, απλώσουν ένα χέρι καλής διάθεση προς τα εθνικά κόμματα και να λάβουν υπόψη όλες τις περιστάσεις ε, που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στο πολιτικό μας περιβάλλον έτσι ώστε οι άνθρωποι στο Συμβούλιο να μην ασχολούνται μόνο με τις θέσεις που είχαν παλιά το 2012 αλλά να προχωρήσουν τώρα για το πώς πάει η αξιολόγηση Ξέρετε κι εσείς πως ο κανονισμός μπήκε σε εφαρμογή το 17. Είχαμε πει το 18 μια έκθεση, αλλά βεβαίως εμείς αυτή τη στιγμή, επειδή έγινε μια έκκληση από το Κοινοβούλιο, είμαστε σε πλήρη ε, δράση έτσι ώστε να προετοιμάσουμε τις απαραίτητες τροπολογίες. Ο κύριος Άνταμ έχει το λόγο. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά. Χρησιμότατη και άκουσα ενδιαφέρουσα συζήτηση και για μας Εμείς δεν συμμετέχουμε σε αυτή την αναθεώρηση, εφαρμόζουμε την ισχύουσα νομοθεσία και θα εφαρμόσουμε τη νέα νομοθεσία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως προανέφερα, αν μπορούμε να βοηθήσουμε με την εμπειρία μας από την πρακτική, με τα χαράς να το κάνουμε. Ήταν πολύ σημαντικό να ακούσουμε όλα τα επιχειρήματα που αναφέρθηκαν. Σύντομα, θέλω να σχολιάσω την ερώτηση του κύριου Μέσου Σμιτ. Δεν ξέρω πώς σχετίζεται με την, αν σχετίζεται περισσότερο με την αναθεώρηση την ισχύουσα την νομοθεσία. Ίσως σε άλλο βήμα θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες. Τόσον αφορά το δικό μας φορέα, ε, εμείς συνεχώς ελέγχουμε κατά πόσο η εκπροσώπηση υφίσταται και πρέπει να ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια καθόλου την περίοδο. Αυτό είναι το σχόλιο που είχα εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου όλων των συναδέλφων μπορώ να πω ότι ήταν εξαιρετικά χρήσιμη η ανταλλαγή απόψεων και για μας και μας είχατε σαφή γραμμή στην απάντηση που δώσατε. Πρέπει η αναθεώρηση να εστιαστεί επί της καλύψεως των κενών που διαπιστώθηκαν και από αυτά που είπε η κυρία Γιώχανσον είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδράζεται επί των άμεσων αλλαγών που απαιτούνται. Αυτό το συμπέρασμα ας συναγάγουμε από αυτή τη συνάντηση και αύριο συνεδρίαση των συντονιστών θα συνεχιστεί η συζήτηση να δούμε αν θα δοθεί συνέχεια και από αυτού με, θα αποφασίσουμε τι πορεία θα ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εκείνους που απεδέχθησαν την πρόσκλησή μας. Ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση. Θα συνεχίσουμε συνάδελφοι. Έχουμε άλλα δύο σημεία στην ημερήσια διάταξή μας. Θα ήθελα λοιπόν να προχωρήσουμε και να πάμε στην γνωμοδότηση του κυρίου Πρέντα. Συνάδελφοι, δεν έχει ολοκληρωθεί συζήτηση, συνεχίζονται οι εργασίες μας. Σας παρακαλώ οι σύμβουλοι να κάνουν λίγη ησυχία. Dan, maybe you try and uh, you see you want to wait a second. Δεν έχω πολύ ισχυρή φωνή, λέει ο κύριος Πέντα. Έχω πρόβλημα με τη φωνή μου. Θα ηρεμήσουν όμως. Θα γίνει ησυχία. Oh. Παρακαλώ αν θέλετε συζητήσεις ε, ιδιαίτερες, όχι εντός εθούς σας παρακαλώ, εκεί στο βάθος. Ο Τέρι Κάμπρας, το είπα το όνομά του. Uh, Συνάδελφοι, σας παρακαλώ Κοιτάξτε, με την ακουστική που έχει η αίθουσα σας ακούμε εδώ. Νομίζετε ψιθυρίζετε, αλλά σας ακούμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρέντα. Πρόκειται περί της δεύτερης ανταλλαγής απόψεων όσον αφορά τη γνωμοδότηση. Έχουμε το κείμενο αυτή τη φορά. Έτσι οι συνάδελφοι μπόρεσαν να σχηματίσουν πιο ξεκάθαρη εικόνα όσον αφορά την κατεύθυνση που ήθελα να δώσω στην γνωμοδότηση. Δεν θα επαναλάβω αυτά που ήδη είπα στην τελευταία ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα να επενθυμίσω όμως σε συντομία κάποια στοιχεία. Πρώτα απ' όλα ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές πρέπει να αλλάξουν, να γίνουν πιο διαφανείς, να έχουν περισσότερο πολιτικό χαρακτήρα. Πρέπει να βρούμε τα μέσα τους ώστε οι πολίτες να αισθανθούν ότι πραγματικά τους ενδιαφέρουν αυτές οι εκλογές, τους αφορούν αυτές οι εκλογές και πιστεύω ο μόνος τρόπος για να καταπολεμήσουμε την αποχή, είδαμε να αυξάνεται η αποχή με την πάροδο των ετών, για να καταπολεμηθεί αυτή η αποχή πρέπει να καταδευτούν προσπάθειες. Κυρίως και οι πρόσφατες ιδέες που προτείναμε, δεν κινητοποίησαν ε, περισσότερο τους πολίτες, αλλά λιγότερο δυστυχώς. Η ιδέα του επικεφαλής του ψηφοδελτίου που θεωρήθηκε σαν, ε, πώς να το πω, εξαιρετικά ελκυστικό, δεν παρήγαγε αποτελέσματα. Το συζητήσαμε αυτό επανειλημμένα άλλωστε. Είμαι στη μειοψηφία, υπάρχει πλειοψηφία συναδέλφων που πιστεύει ότι αυτό είναι μια καλή ιδέα. Ίσως είναι μια καλή ιδέα, αλλά όχι για την αύξηση της συμμετοχής στις εκλογές. Για την ώρα δεν έδωσε αποτελέσματα. Πιστεύω ότι σε κάποια χρόνια θα βλέπουμε πιο ξεκάθαρα. Δεύτερο σημαντικό, ουσιαστικό σημείο, Δεύτερο σημείο σημαντικό, πρέπει να έχουμε διάβια πνεύματος. Μας αρέσει να κάνουμε καλές ομιλίες και να δημιουργούμε ουτοπικές ιδέες, ο καθένας στην ομάδα του, αλλά εγώ βλέπω τα πράγματα ως έχουν, με μακιαβελικό τρόπο. Δεύτερο, οι πρωτοβουλίες, οι, των πολιτών, οι ευρωπαϊκές, υπάρχει συνένεση, συμφωνία, άποψη στο Κοινοβούλιο. Προσωπικά ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί ο κανονισμός και έτσι οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν με αποτελεσματικό και ικανοποιητικό τρόπο να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο της πρωτοβουλίας των πολιτών. Τρίτον, η ασφάλεια, μία από τις βασικές ε, ανησυχίες των πολιτών, θα πρέπει ο ρόλος που παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια των Ευρωπαίων να υπογραμμιστεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα έκανε πολλά για να ετοιμάσει θεματολόγιο την ασφάλεια θα πρέπει κατά την άποψή μου τα κράτη-μέλη πλέον να παίξουν το παιχνίδι και ε, να φροντίσουν να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών και να υπάρχει η διαλειτουργικότητά τους. Στην πρώτη συνάντηση είπα ότι το Brexit και οι συνέπειες για τα δικαιώματα των Βρετανών πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών πρέπει να συμπεριληφθεί στη γνωμοδότηση. Και η θέση της κ. Τερέζα Μέη δεν είναι καθυσυχαστική. Παρά τις δηλώσεις των Βρετανών οι προτάσεις που υπέβαλε δεν δίνουν καμία ασφάλεια και βεβαιότητα για το μέλλον. Θα πρέπει να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, πάση θυσία, και δεν μπορούμε να κυρώσουμε ε, ε, καμία συμφωνία που τους κάνει πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Με την πάροδο του χρόνου βλέπουμε ότι επικρατεί μεγαλύτερη αβεβαιότητα παρά βεβαιότητα και σαφήνεια σχετικά με αυτά που πρόκειται να συμβούν. Εγώ πιστεύω, αν θα έχουμε το φθινόπωρο μεγαλύτερη σαφήνεια. Εγώ πιστεύω ότι συνεχώς ε, χειροτερεύει η κατάσταση. Και ε, πιστεύω ότι τρέφονται αυταπάτε ε, σύμφωνα τι οποίε με το Brexit έχουμε καλύτερη συμφωνία από ό,τι είχαμε πριν με τη συμφωνία του Κάμερον εν ώψη του δημοψηφίσματο. Εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι μεγάλη αυταπάτη. Ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε μετά την ψήφο των Βρετανών περισσότερα από αυτά που είχαμε πετύχει συμφωνία με τον Κάμερον. Αυτό δεν κατάλαβα γιατί το πιστεύουμε. Γιατί το τροφοδοτούμε αυτό. Α, ε, αυτή τη φαντασίωση. Έχουμε διαπραγματευτές βέβαια και έχουμε μια ομάδα που ασχολείται με το θέμα των διαπραγματεύσεων. Τώρα κατά την ταπεινή μου, για την γνωμοδότησή είμαι 6 Σεπτεμβρίου είναι η ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών. Εγώ θα δώσω κάποια στοιχεία όσον αφορά την προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεως στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Εκεί έχει μπλοκαριστεί εδώ και αρκετά χρόνια. Στην προηγούμενη θητεία για την Επιτροπή, υποεπιτροπή ε, ε, την νομική είχα ετοιμάσει κάποια γνωμοδότηση την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Θα πρέπει να γίνει πρόοδο στο Κοινοβούλιο, να πιέσει για πρόοδο αυτό το θέμα, διότι αυτή η προσχώρηση τη Ένωση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν είναι μόνο νομική υποχρέωση, αλλά θα επέτρεπε και καλύτερη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Προσωπικά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα συνεκτικό σύστημα για την προστασία των δικαιωμάτων στην Ευρώπη είναι και θέμα αξιοπιστίας που τίθεται της εξωτερικής μας πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την πολιτική της διεύρυνσης και θα πρέπει να ζητούμε από τις υποψήφιες χώρες να ακυρώνουν τη σύμβαση αλλά ε, δεν, υπάρχει, ε, ε, δεν υπάρχει εποπτεία της ενώσεως όμως από την άλλη και των κρατών μελών αυτής από τις αρχές της αρμόδιας της συμβάσεως. Πρέπει να σταματήσει αυτή η παράλογη κατάσταση πολιτικός παράδοξη αυτή η κατάσταση που ανέφερα. Ελπίζω οι συνάδελφοι να συμβάλλουν στη διατύπωση νομοδοτήσεως και θα εθετήσουμε τελικά ένα κείμενο το οποίο θα έχει προστιθέμενη αξία, θα δώσει προστιθέμενη αξία από τον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κλάουντια Ταπαρντέλ έχει το λόγο για τους ελιστές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την παρουσίαση της θέσης του. Και εμείς Ελπίζουμε ότι οι συζητήσει θα οδηγήσουν μια καλή γνωμοδότηση. Η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών είναι, είναι πολύ σωστή. Όπως ε, αναφέρθηκε και προηγουμένω στι 20 Ιουνίου, πιστεύουμε ότι όπως είπα και στις 20 Ιουνίου, πιστεύω ότι αυτή η έκθεση και αυτή η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας είναι πολύ σημαντικά στοιχεία θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι οι πολίτες θα μπορούν να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους όταν εργάζονται, ταξιδεύουν, ε, σπουδάζουν ή συμμετέχουν στις εκλογές ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και θα πρέπει να στερνίζονται τις κοινέ αξίες οι πολίτες. Αυτό που με προβληματίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι οι πολλοί Ευρωπαίοι ακόμα δεν έχουν επίγνωση των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν στους Ευρωπαίοι πολίτες. Αναφέρομαι στα δικαιώματα για τις εκλογές ή για την ε, ε, προστασία που παρέχουν οι προξενικές αρχές σε άλλα κράτη-μέλη. Και υπήρξε πολύ χαμηλή συμμετοχή στις ευρωεκλογές τα τελευταία χρόνια ε, αυτό διαπιστώσαμε. Ε, η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ χαμηλή, κυρίως ε, στους νέους. Πολλοί από τους νέους παραδέχονται ότι δεν είναι ενήμεροι για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και κατά πώς συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη βελτίωση της καθημερινής τους ζωής. Και αυτό πρέπει να είναι ένα μήνυμα συναγερμού για μας ε, θα πρέπει οι συστάσεις Επιτροπής ΑΦΚΟ να επικεντρωθούν στην επίλυση των προβλημάτων με μια σύντομη προθεσμία, δηλαδή να, βρεθούν, να λυθούν τα προβλήματα πριν τις εκλογές του 2019 και πριν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το Brexit. Ε, μπορούμε να πούμε ότι περάσαμε πολλά χρόνια κρίσεως, αλλά η μεγαλύτερη τέτοια κρίση ξέσπασε με την ε, ενεργοποίηση του άθρου 50 για το Brexit θα πρέπει να καθορίσουμε λοιπόν σωστές προτεραιότητες και να λάβουμε σοφές αποφάσεις υπέρ των πολιτών. Χαίρομαι διότι στη γνωμοδότησή του κ. Πρέντα τονίζει τη σημασία που έχει η πρωτοβουλία των πολιτών. Χρειάζεται ένα εργαλείο για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στην Ευρώπη μετά την αξιολόγηση της εφαρμογής αυτή τη πρωτοβουλία των πολιτών από τη θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα, πιστεύουμε ότι μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται μια αναθεώρηση του μέσου αυτού και ελπίζω ότι θα ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του εργαλείου αυτού μέχρι το τέλος ε, του τέχοντο έτους. Τώρα όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών των πολιτών και ποια είναι η εμπιστοσύνη που έχουν οι πολίτες όσον αφορά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οι πολίτες περιμένουν να καταπολεμά με πιο ενεργό τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση την τρομοκρατία. Είδαμε διάφορες απόπειρες, πολλές επιθέσεις οι οποίες έλαβαν χώρα τα τελευταία δύο και τρία χρόνια. Ε, πιστεύω ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να συντονίζει καλύτερα τις εσωτερικές και εξωτερικές δράσεις της για την ασφάλεια για να προστατεύει καλύτερα τους πολίτες. Όμως, εγώ διστάζω κάπως ε, όσον αφορά το κατά πόσο η πολιτική ασφαλείας και της μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα πρέπει να αποτελεί ένα κομμάτι αυτού του ζητήματος που ζητούμε τώρα. Συμφωνώ με τις περισσότερες από τις προτάσεις του κ. Πρέντα κατά τα άλλα και βεβαίως θα εκφράσουμε συγκεκριμένη θέση εμείς σαν ομάδα σοσιαλιστών στις τροπολογίες που θα υποβληθούν. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον να θέλει να μιλήσει στους φιλελεύθερους. Για τους πράσινους ο Τέρι έχει κάτι να πει. Γερμανικά, από ό,τι καταλαβαίνω. Αγγλικά, αγγλικά σας αρέσουν. Ωραία διότι δεν είναι δυνατό να μιλήσω καταλανικά. Θα ήθελα να μιλήσω καταλανικά, αλλά δεν μπορώ. Αν πληρώσετε μπορείτε, λέει η Πρόεδρος. Ε, καλώς. Υπάρχουν ένα-δύο πράγματα που θα ήθελα να πω, ένα-δύο σημεία που υποστηρίζουμε και ένθερμα στην πρόταση του συγγητού, συγκεκριμένα την ανάγκη μεταρρύθμισης ε, του συστήματος καταχώρησης που θα είναι λιγότερο ε, ε, περιοριστικό όσον αφορά τι ευρωπαϊκέ πρωτοβουλίε πολιτών, να πλουστευτεί η διαδικασία συλλογή υπογραφών και να δίδεται σωστή συνέχεια σε κάθε επιτυχή πρωτοβουλία. Ξέρει και ο κ. Σέφλιν, αυτό, αυτή είναι η βασική μου ιδέα. Είναι πολύ καλό να συμβαίνει κανείς όταν συλλέξει κανείς ε, ένα εκατομμύριο υπογραφές, αν δεν συμβαίνει τίποτα, είναι ένα παιχνίδι και πάρα πολύ δαπανηρό μάλιστα. Μετά υποστηρίζουμε και την ε, προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών που θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες διαπραγματεύσεις για το Brexit. Όμως υπάρχει ένα σημείο που θα τονίσω. Στην πρόταση του εισηγητού για την ασφάλεια δεν γίνεται καμία αναφορά στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτό. Ξέρω ότι θέλετε να τα σέβεστε, είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά θα έπρεπε να αναφέρετε ρητά διότι αυτό είναι κρίσιμο σημείο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα από το e Α, η Μπάρμπαρα, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την εργασία του και υπάρχουν σημεία σύγκλησης ιδιαίτερα για τη δυνατότητα τροποποίηση του εκλογικού νόμου και για τις ε, βρετανικές για διαπραγματεύσεις με τον Brexit για τα δικαιώματα των πολιτών και για την αναθεώρηση της πρωτοβουλίας των πολιτών. Για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών. Βεβαίως συμφωνώ να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των ε, πολιτών. Αλλά υπάρχει μία απόφαση του δικαστηρίου για την πρωτοβουλία για το TTIP και για τα δικαιώματα κάποιων μειονοτήτων αποδείχθηκε ότι η Επιτροπή δεν τα προώθησε αλλά αντίθετα προσπάθησε να τα περιορίσει και έδειξε απροθυμία. Βεβαίω πρέπει να αυξηθούν οι προσπάθειε για την πρόθεση αυτών των δικαιωμάτων. Και πρώτα απ' όλα οι ρήτρε αυτέ θα πρέπει να μπουν στι συνθήκε ή σε μια χάρτα των ανθρωπίνων, μια νέα χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε κάτι νέο, αλλά απλώ να εφαρμόσουμε αυτό που ήδη υπάρχει στο πρωτογενέ ενωσιακό δίκαιο για τον ίδιο λόγο. Συμφωνεί απόλυτα με το δεύτερο τμήμα της πρώτης παραγράφου ότι πρέπει να υπάρχει σαφής δέσμευση από κράτη-μέλη. Αυτός δεν είναι ο μόνος τρόπος για να προστατευτούν τα δικαιώματα των πολιτών. Έχουμε μια σειρά από κοινού και δεσμευτικούς κανόνες για το σκοπό αυτό και πρέπει να τους ε, αξιοποιήσουμε πλήρως. Σημειώνω ότι ούτε η έκθεση της Επιτροπής, ούτε η γνωμοδότηση εδώ αναφέρονται στην Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Νομίζω ότι από πλευρά ΑΦΚΟ είναι σημαντικό να αναφερθούμε στη Χάρτα. Τώρα κάποια άλλα σημεία. Στην παράγραφο 2. Συμφωνώ με τον εισηγητή. Ο εκλογικός νόμος πρέπει να βελτιωθεί και να γίνει πιο διαφανής. Όμως η διαφάνεια και η συμμετοχή δεν πρέπει να είναι μόνο κατά τη στιγμή των εκλογών. Οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν συνεχώς. Όπως βλέπουμε με τα κινήματα κατά της διαφθοράς των πολιτών. Υπάρχει διάθεση δηλαδή. Καθώς και στις ε, προσφυγές των ε, Ευρωπαίων διαμεσολαβητή. Οι περισσότερες προσφυγές αφορούν την έλλειψη διαφάνειας, ιδιαίτερα σε θέματα οικονομικής πολιτικής στην παράγραφο 3 την οποία χαιρετίζω αλλά ίσως θα την ενίσχυα και θα ήθελα να συνδυάζεται καλύτερα με αυτά που είπατε εσείς για τις ε, προτάσεις της κυρίας Μέη. Λέτε ότι πρέπει κάποια θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να προστατευτούν από τη Συμφωνία Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί. Να αναφερθούμε στο σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εννοησιακή υπηκότητα και την ελεύθερη κυκλοφορία. Όλα αυτά πρέπει να προστατευτούν. Περαιτέρω. Κατά τη γνώμη μου, η Συμφωνία για τα Δικαιώματα των Πολιτών πρέπει να αντιμετωπιστεί και χωρισμένα από οποιαδήποτε άλλα τμήματα της διαπραγμάτευσης. Ξέρω ότι δεν είναι αυτή η άποψη του κυρίου Φερχόφστατ. Αλλά πρέπει να πω ότι ελπίζω ότι η κυρία Χιούμπνερ θα παρουσιάσει στις συζητήσεις ε, στην ομάδα για τον Brexit και τις άλλες απόψεις για το πόσο πρέπει να αντιμετωπιστεί χωριστά το θέμα των δικαιωμάτων των πολιτών. Παράγραφος 4. Θα συζητήσουμε την πρωτοβουλία των πολιτών πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια της έκθεσης Σέπφλιν. Όπως είπα, θα ήμουν πιο επιφυλακτική έναντι του σχεδίου της ε, Κομισιόν που είναι κυρίως ε, τεχνικής φύσης τροποποίηση. Μετά την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου πρέπει να γίνει πραγματική αλλαγή πορείας στη διαδικασία αποτίμησης. Τέλος παράγραφος 5. Ειλικρινά δεν μπορώ να πω ότι με συναρπάζει. Η ασφάλεια είναι προτεραιότητα. Αλλά όχι η πρώτη προτεραιότητα. Η η ηθαγένεια και η συμμετοχή στα κοινά και η αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού αποχής. Όλα αυτά συνδέονται απευθεία με την ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη των πολιτών. Σημαίνει πως θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι, να υπάρχει ένταξη όλων στην κοινωνία, να υπάρχει ελεύθερη συζήτηση και να προβλέπονται η κάλυψη των βασικών αναγκών των πολιτών. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν πλήρως στη δημοκρατική ζωή. Αυτές οι αρχές λυπάμαι, αλλά δεν υπάρχουν στο κείμενο, αλλά θα τις προτείνω μέσω τροπολογιών. Θέλετε να κάνετε σχόλια, George, θες κάτι να πεις? Βεβαίως. Τρία λεπτά. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία ε, πυροδότησε μία σειρά από που θα ήθελα να προσθέσω. Αν καταρχήν μιλάμε για δικαιώματα πολιτών, να σας πω πως ο τρόπος να τα στηρίξουμε είναι μια συνεχής επαφή με τους θεσμούς, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς εδώ. Δηλαδή, πώς μπορεί ένας πολίτης να έρθει σε επαφή με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είναι εξαιρετικά περίπλοκο, πολύ δύσκολο και κυρίως ε, γιατί έχουμε αυτή τη δι, διτή ηθαγένεια. Γιατί οι περισσότεροι από τους... Ε, ε, συμπολίτες μου γνωρίζουν ότι είναι Ούγγροι πολίτες, αλλά δεν ξέρουν ότι είναι ε, Ευρωπαίοι πολίτες και θυμόσαστε ε, το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία. Υπάρχει ένα είδος ε, απόζευξης μεταξύ των δύο και αυτό πρέπει να το ξεπεράσουμε, αποσύνδεσης. Ε, δεν είναι ίσως εδώ ο κατάλληλος τόπος και νομίζω ότι από το 9 μέχρι 14 είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξελίχθηκε, αλλά η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλεγές ε, καθ' όλη την πορεία του δημοκρατικού κόσμου μειώνεται συνέχεια. Και αυτό έχει να κάνει με την κοινωνία των πολιτών. Δηλαδή δεν είναι πια ο νομοθέτης ο οποίος έχει μόνο την εξουσία πριν από 30-40 χρόνια. Έχουμε το ΜΚΟ, έχουμε την κοινωνία των πολιτών και άλλους τρόπους για να έρχεται κανεί σε επαφή με την εξουσία. Οπότε όταν τα σκέφτεσαι όλα αυτά, σκεφτείτε ότι μπορεί να έχουμε και ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών που δεν λειτουργεί μόνο στις Βρυξέλλες όπου συγκεντρώνεται, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ή θα έπρεπε να υπάρχει και σε όλες τις εθνικές πρωτεύουσε. Συνάδελφε, η συζήτηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ξέρω πως στην εποχή αυτή Ακόμα πιστεύουμε πως η καλή δημοκρατία, το καλό καθεστώς γενικότερα ε, αποδεικνύεται από υψηλή συμμετοχή. Δεν ήταν πάντα έτσι. Και όπως είπε ο συνάδελφος ε, Σόπλινγκ μόλις, τα τελευταία χρόνια είδαμε διαφορετικού είδους κινητοποιήσεις από την κοινωνία των πολιτών, όχι μόνο από τους εκλογείς. Γιατί οι πολίτες έχουν το δικαίωμα ψήφου, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο είναι ενδιαφέρον και δεν ξέρω αν αυτές τις ιδέες μπορούμε να τις πλαισιώσουμε περισσότερο αναφερόμενοι στην κινητοποίηση των ε, εκλογέων, συγκινητοποίηση των πολιτών και αν θεωρούμε πως, πια, πως αυτή είναι η καλή πολιτική κοινότητα, ε, έτσι όπως ε, λέγαμε στο παρελθόν. Εγώ θέλω να ευχηθώ καλές διακοπές σε όλους τους συναδέλφους και να σας πω πως εγώ στις διακοπές μου θα γράφω τροπολογίες. Στα γρήγορα να σας υπενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα για την έκθεση. Σήμερα τη συστήσαμε τη γνωμοδότηση. Προθεσμία για τροπολογίες 6 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα. Και μετά, 28 Σεπτεμβρίου, θα γίνει στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων η σχετική ψηφοφορία. Η Μπάρμπαρα έφυγε. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στο τελευταίο σημείο της ημέρης διάταξης που είναι το πολιετές ε, χρηματοδοτικό πλαίσιο να προετοιμάσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου για, το, ε, για τη μετά το 2020 εποχή. Ο κύριος Άνεμανς έχει το λόγο. Ξέρετε πως πέρσι είχα την τιμή να προετοιμάσω ένα σχέδιο γνωμοδότησης για την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα θέμα το οποίο ε, δυστυχώς κατέληξε άσχημα μια και απερίφθη το κείμενό μου ακριβώ επειδή το έγραψα εγώ. Αλλά εγώ δεν θα αλλάξω. Δεν θα αλλάξω στρατηγική. Εγώ ανεξάρτητα με τις προσωπικές μου υποθέσεις πάντα συντάσσω κείμενα όσο μπορώ πιο πολύ αντικειμενικά. Και να σας πω πως στο πρώτο σημείο τονίζω πως ο διάλογος μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου θα πρέπει να ενισχυθεί και θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια διαδικασία που θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του προγράμματος και όχι να επιβληθεί μια ε, διαδικασία από την κορυφή προς τη βάση όπως κάνει συνήθως το Κοινοβούλιο. Τώρα θα γυρίζω στα Ολλανδικά για να πω τα υπόλοιπα όπως κάνω συνήθως και να σας πω πως νομίζω ότι στο κείμενό μου αποδεικνύω πως έχω τη δυνατότητα να αφήσω στην άκρη τις προσωπικές μου απόψεις και να ασχοληθώ με το θέμα αντικειμενικά. Τώρα, μιλώ για το θέμα της ομοφωνίας και για το κατά πόσο μπορούμε να μετακινηθούμε προς μια ειδική πλειοψηφία και για το σημείο 4 να σας πω πως και πάλι αφήνω στην άκρη τις προσωπικές μου απόψεις και λέω πως δεν συμμορφούνται το σημείο αυτό με τις συνθήκες, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να λαμβάνει αποφάσεις για τις διαπραγματεύσεις ε, εκεί που δεν έχει αρμοδιότητα. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να προσπαθεί να επεκτείνει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Συμβούλου εκεί που δεν υπάρχουν. Και νομίζω ότι αποδεικνύω την καλή μου θέληση όταν μιλώ για τις ευρωπαϊκές αρχές Και να σας πω πως υπάρχει ε, στο επόμενο θέμα και μια δυνατότητα εξοικονόμησης πόρων σε εθνικό επίπεδο για, ε, ε, στα πλαίσια των μελλοντικών χρηματοδοτήσεων και μετά ε, λέω πως θα πρέπει να προσαρμοστούμε ε, στη χρηματοδότηση έτσι ώστε η αποφάση που παίρνουμε να συμπίπτει ε, με την περίοδο χρηματοδότησης. Τι σημαίνει αυτό με άλλα λόγια. Θα πρέπει οι δημοσιονομικές προοπτικές να μην είναι επταετής όταν ψηφίζονται, αλλά πενταετής, άρα να τρέχουν παράλληλα με τη θητεία μας. Τώρα, μετά, συνέπειες του Brexit, κάτι το οποίο συζητήσαμε σήμερα το πρωί, όλοι γνωρίζουμε πώς θα γύρει μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Όλοι ξέρουμε πως θα είναι δύσκολο να προβλέψουμε τις ε, συνέπειες του Brexit και για το επόμενο ε, πολιετές πρόγραμμα δεν θα είναι καθόλου εύκολο να μαντέψουμε τι θα χρειαστεί. Και αυτό θα πρέπει να ακουστεί γιατί είδαμε και το θέμα των διαπραγματεύσεων και πόσο σαφή είναι τόσα ζητήματα. Υπάρχει κάποιος ο οποίο θα ήθελε να σχολιάσει από το ΕΛΚ ή από τους σοσιαλιστές. Κυρία Μπρέσο. Δεν βλέπω από το ΕΛΚ. Ορίστε, είμαι σκιώδη, λέει κύριε Μπρέσο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για τη δουλειά που έκανε Βλέπω και εγώ ότι κατέβαλε μια προσπάθεια δικημενικότητας. Ασύνηθες στην ομάδα του. Όχι πάντα από τον ίδιο. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν λοιπόν για να μην συμβεί αυτό που μας υπενθύμησε. Διότι οι σχέσεις μεταξύ των ομάδων μας δεν είναι καλές. Θα ήθελα να υπογραμμίσω μόνο κάποια πράγματα. Και μετά θα υποβάλουμε τροπολογίες επί των σημείων εκείνων επί των οποίων έχουμε αμφιβολίες. Καταρχάς, πάνω απ' όλο πιστεύω ότι δεν είναι αποδεκτό στο σημείο 5, το σημείο 5 δεν είναι αποδεκτή η ιδέα από το Brexit να οδηγηθούμε σε μείωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Σίγουρα θα επιφέρει μία μείωση που οφείλεται στην έλλειψη της συνεισφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα αντισταθμιστεί προφανώς από μερική μείωση των χρημάτων που λαμβάνει τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως η συζήτηση για το μελλοντικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους πόρους μας δείχνει ότι κάτι συζητείται. Να βρεθούν οι ίδιοι πόροι, ε, ε, τώρα πώς θα βγουν από τους εθνικούς προϋπολογισμούς που υποφέρουν. Είναι δύσκολο να ζητήσουμε θυσίες από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. αλλά μέσω αναπτύξεως ιδίων πόρων και εξαλείφοντας τις επιστροφές, rebates, σε όλους και όχι μόνο αυτά που αναλογούν στη Μεγάλη Βρετανία. Πράγματα που αναφέρονται και στην έκθεση Verhofstadt και στη δική μας. Το θέμα των πόρων είναι ανοιχτό και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να επενθυμιστεί κυρίως από μια επιτροπή όπως των συνταγματικών υποθέσεων ότι τα 410 και 311 των συνθήκων αναφέρουν ότι νέες πολιτικές και νέες δραστηριότητες συνεπάγονται και τη διάθεση επαρκών πόρων για τις δραστηριότητες αυτές. Πρέπει να υπάρχει συντισμός μεταξύ δραστηριότητες και πόρων. Οι δραστηριότητες έχουν αυξηθεί πολύ, εξακολουθούν να αυξάνονται, υποβάλλονται νέες προτάσεις για στόχους, άρα σκόπιμο θα ήταν να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την έννοια των ε, συνθήκων θα πρέπει οι πόροι που διατίθεται να αντιστοιχούν στα καθήκοντα. Αν θέλουμε να κάνουμε σε κάποια πεδία περισσότερα πράγματα πρέπει να βρούμε νέους πόρους για να διατεθούν, για να καλυφθούν οι νέοι τομείς. Δεύτερον, όπως αναφέρθηκε και από το έγγραφο για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, θα πρέπει να διερευνήσουμε και την ιδέα του να συνδέσουμε την εκταμείωση των πόρων από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, όχι σύμφωνα με τους κανόνες του προπολογισμού μόνο, αλλά και ε, ανάλογα με το, με το κράτος δικαίου στα κράτη-μέλη παραβιάσεις των ευρωπαϊκών κανόνων. Τώρα πια δεν είναι... Ε, δεν συνδέονται μόνο με, την, ε, με, τους κανόνες του προπολογισμού, αλλά σχετίζονται και με το μη σεβασμό των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και, των κανόνων ε, που σχετίζονται φερρυπίν με διάφορα θέματα όπως είναι αυτό των μεταναστών. Στο σημείο 3 συμφωνούμε ότι πρέπει να μειωθεί ο χρόνος του πολίτη του δημοσιονομικού πλαίσιου από 7 χρόνια, η διάρκεια του να είναι 5 χρόνια, αλλά να μιλάμε 5 συν 5, διότι όπως γνωρίζετε για κάποια προγράμματα όπως η πολιτική συνοχή στα 5 χρόνια είναι πολύ σύντομη περίοδος, άρα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Μείωση ναι, αλλά να επενθυμίσουμε και την περίπτωση 5 συν 5 με πλήρη αναθεώρηση ενδιάμεση στα 5 χρόνια. Ιδού αυτά είναι κάποιες σκέψεις Βέβαια επιφελεσόμαθα να υποβάλουμε τροπολογίες και θα αξιολογήσουμε τη θέση μας στην ψηφοφορία μετά από τη συζήτηση που θα γίνει για και την ψηφοφορία της τροπολογίας. Ευχαριστώ. Ελκ, Ράντζελ, ε, κανένας από τους άλλους σκιώδες δεν είναι παρόν. Ελπίζω όμως να έρθει σε επαφή μαζί τους για τη συνάντηση των σκιωδών. Θέλετε να κλείσετε κύριε Γκέροντ. Ευχαριστώ την κυρία Μπρέσο για την αντίδρασή της. Θα επιχειρήσω να λάβω υπόψη τα θέματα που ανέφερε. Πρέπει να τονίσω ότι ναι μεν έχουν συνεργαστεί πολύ καλά οι ομάδες μας στο παρελθόν, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας αποτρέψει από το να το επιδιώξουμε. Μπορεί να διαχωρίσω το ρόλο του εισηγητή από τις απόψεις που θα δω τι μπορώ να κάνω θα προσπαθήσω να συντάξω μια έκθεση που να τύχει ευρεία στηρίξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και η Πρόεδρος. Να σε ενημερώσω για τις προθεσμίες, για το θέμα αυτό. Προθεσμία για τροπολογίε η 6 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα. 6 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες 28 Ενάτου και ελπίζω να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 11 Οκτωβρίου και σας διαβεβαιώ ότι η Γραμματεία μπορεί να σας βοηθήσει για να ε, εκπονήσετε συμβαστικές τροπολογίες σε ένα μεταγενέστερο στάδιο. Είμαστε στη διάθεσή σας. Λοιπόν, διάφορα. Δεν έχω τίποτα στα διάφορα. Επόμενη συνεδρίαση στις 4 Σεπτεμβρίου το απόγευμα στις 3. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση σε όλους. Τα ξαναλέμε τον Σεπτέμβριο. Και δυστυχώς όμως η συνεδρία των συντονιστών υπάρχει ακόμη αύριο πρωί. Ευχαριστώ πολύ.